μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας και να ελπίσουμε ότι θα έλθουν και άλλοι συνάδελφοι μαζί μας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ ησυχία, ησυχία και στην είσοδο και ξεκινώντας ε, αλλαγή των σημείων 6 ε, και 7 της ημερησίας διάταξης ε, μετά από την αρχή και τα τυπικά θα έχουμε ε, θα στο 7 για το Πακιστάν την αποστολή και μετά το επόμενο για τα φράγματα και έτσι ορισμένοι μέλη που θα ήρθαν εδώ θα είναι παρόντα για αυτή τη συζήτηση. Μήπως για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης γιατί για τη μέση διάταξη υπάρχει κάποια αντίρρηση. Όχι. Αλλάζει λοιπόν η ημερήσια διάταξη και ισχύει. Έτσι. Έχετε τα πρακτικά συναντρίες 3 Μαρτίου. Αν έχετε κάποιο σχόλιο πριν από τη συναντησή μα σήμερα μπορείτε να το πείτε στη γραμματεία διαφορετικά θα εγκριθούν αυτά τα πρακτικά. Προηγουμένω λοιπόν είπαμε το 7 πρώτα και το 6 δεύτερο. Ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε, μάλλον ώρα των ερωτήσεων δύο, μία της κυρίας Κέλλερ για το πλαίσιο το αυτές και της κ. Πατίνη για την πράσινη βίβλο για την ε, πολιτική ανάπτυξη τη μελλοντική Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές, θα έχουμε, αυτές ερωτήσεις έχουμε σε γαλλικά και αγγλικά. Ξεκινάμε με το ερώτημα της κυρίας Κέλλερ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Μήπως μπορεί να δώσει μια απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, δεν βλέπω και καλά με αυτά τα γυαλιά. Θα πρέπει να συνηθίσω να έχει το λόγο κυρία μου. Έχετε το λόγο κυρία Μπουλγκάτ. Ναι, σας ευχαριστώ. Και να χαιρετήσω όλους. Μια ερώτηση για το πολιετές πλαίσιο το οικονομικό και αυτό που ακούστηκε από πλευράς Επιτρόπου Μέλστρομ για τις θετικές προτάσεις. Να υπενθυμίσω πως έχει το πλαίσιο του θέματος. Όχι που γνωρίζετε. Εντάξει. Στη Γενική Διασύντευκο ενημερωθήκαμε για την πρόταση αυτή Μέλστρομ και είχαμε και αρκετές επαφές σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Η Γενική αυτή δεν μας υπέβαλε καμία λεπτομέρεια πρόταση για να δούμε ακριβώς το τι ακριβώς θα ήθελε να χρηματοδοτήσει στα πλαίσια αυτής της πρότασης και συνεχίζουμε τις επαφές μαζί τους τώρα. Όπως έχει όμως η κατάσταση Η τάση της πρότασής μας είναι να βοηθήσει την πρόταση της Digihome, αλλά υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Εντάξει, μπορούμε να δεχτούμε η Γενική Αυτή με το νέο δημοσιονομικό της εργαλείο να το χρηματοδοτήσει από το κεφάλαιο 3 της ε, δράσης σε τρίτες χώρες και βάσει όμως τριών βασικών κριτηρίων απαραίτητων, ε, δεν είναι αποκλειστικά αυτά, θα πρέπει να ισχύουν παράλληλα να ανταποκρίνονται στο συμφέρον και στον τομέα αυτό που ασχολείται η Ένωση με την εντολή συνετάμεσα της ε, Γενικής και να είναι βραχή πρόθεσμες δράσεις να μην είναι δημοσία βοήθεια στην ανάπτυξη στα πλαίσια του ορισμού του ΩΣΑ. Να σας πω κάτι από δικής μας πλευράς. Διαφωνούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει εις βάρος ε, των δημοσιονομικών εργαλείων του κεφαλού 4 με τομιακά σημεία. Αυτό το θέμα της μετανάστευσης είναι κάτι το πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ανάπτυξης και δεν είναι αυτές οι ενέργειες που ανταποκρίνονται στα τρία κριτήρια που αναφέρθηκαν, δεν είναι στα πλαίσια είναι εξωτερικέ συνεργασία, αλλά όχι ανάπτυξη. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε μια παρόμοια μεταφορά κονδυλίων προς την Γενική Δευσίγων. Από δική μας πλευρά θα πρέπει πλαίσια του κεφαλαίου 4 να διατηρηθούν για τη μετανάστευση και το άσυλο γιατί καλύπτουν ενέργειες ε, μεσοπρόθεσμες και, βραχο... μακροπρόθεσμες ε, που είναι ενέργειες ανάπτυξης. Νομίζω ότι απάντησα έτσι. Αν θέλετε κάτι να διευκρινίσω περαιτέρω είμαι στη διάθεσή σας. Ναι, μπορείτε να μας πείτε και γραπτός να μας τα... τα αυτά. Ναι, σίγουρα. Κύριε Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Απλώ για να καταλάβω καλά. Μα λέτε ότι δεν θα σα πείραζε ή θα συμφωνούσατε, εν πάση στην πρόταση της Ρόμ να ε, υπάρχει για την επανεισδοχή ε, κάποια κεφάλαια, αρκεί να είναι τα δικά της ε, χρήματα και όχι αναπτυξιακά κεφάλαια. Και ε, σε βαθμό, που, στο βαθμό βέβαια που δεν πηγαίνουν σε εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας είπατε αν κατάλαβα καλά. Εξαρτάται. Εξαρτάται τι εννοούμε χρηματοδότηση των συμφωνιών επανεισδοχής και επαναπατρισμού. Γιατί εάν υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής στο πρώτο σημείο που ανέφερα, μιλάμε για την παρέμβαση στις τρίτες χώρες, είναι καινούριο, δεν διαφωνούμε, αρκεί να πληρούνται αυτά τα τρία κριτήρια. Τώρα, όταν μιλάμε για τις συμφωνίες επανεισδοχής, χρειαζόμαστε κονδύλια, αλλά το πρόβλημα που υπάρχει είναι η επανεισδοχή ε, σε χω... Ε, από χώρες που είναι διαφορετικές από τις χώρες τις οποίες επαναπατρίζουμε κάποια άτομα. Δηλαδή, αν θέλετε να επιστρέψει κάποιο στη χώρα του είναι ένα θέμα, αλλά αν θέλετε να πληρώσετε για να φύγει κάποιο από την, ε, από την Αίγυπτο και να γυρίσει, για παράδειγμα, όχι στην Ιγυρία, αλλά ε, στην Ερυθρέα, είναι ανάπτυξη. Αν όμως πρόκειται για χρηματοδότηση συμφωνιών ε, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργάνων τρίτων χωρών για την ανάπτυξη υποδομών και για τη διευκόλυνση του καλύτερου χειρισμού ε, της ε, ενσωμάτωσης των μεταναστών ε, στις χώρες προέλευσής τους, αυτό επίσης είναι μία αναπτυξιακή βοήθεια. Εκεί δεν συμφωνούμε. Οπότε λοιπόν εξαρτάται από το τι θα πει αγορά συμφωνιών επανεισδοχής. Νομίζω ότι ο ορισμός των κριτηρίων που αναφέραμε ανταποκρίνονται σε ένα άμεσο ε, συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βραχυπρόθεσμο ε, και ε, νομίζω ότι αυτό αποτελεί ήδη ένα στοιχείο απάντησης. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο ερώτημα της κυρίας Αργεντίνη. Πάλι θα έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος απαντάει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική, το πρώτο ερώτημα αφορούσε το αντίκτυπο των επενδύσεων που μπορεί να έχει αυτό στο, στα στόχους ενέργειας και ανάπτυξης ευρωπαϊκής πολιτικής και θέλουμε να τονίσουμε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνονται στην αηφόρο ανάπτυξη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή ε, που γίνονται και σε επίπεδο ΟΗΕ. Προσπαθούμε πάρα πολύ να προωθήσουμε τις διαδικασίες χαμηλών εκπομπών αερίων για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων και θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτό σε αυτήν την μέγιστη αύξηση δύο βαθμών ε, Κελσίου ε, της ε, θερμοκρασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει πάρα πολλά προγράμματα και σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική αλλά και σε κάθε χώρα ξεχωριστά και καμία από τις επενδύσεις αυτές δεν έχουν κατά τη γνώμη μας συμπεριληφθεί σε αναπτυξιακή βοήθεια. Αντιθέτως, μάλιστα. Τώρα, σε επίπεδο τώρα διεθνές, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, νομίζουμε ότι κινούμεθα προς μια συμφωνία, ε, ε μια παγκόσμια συμφωνία κλιματικής αλλαγής. Αν γίνει κάτι τέτοιο στους επόμενους μήνες, το γεγονός ότι θα ληφθεί υπόψη η τιμή του άνθρακα σε όλες τις διαπραγματεύσεις και σε επενδύσεις, ε, θα σημαίνει ότι από οικονομική απόψεως οι επενδύσεις αυτές θα είναι πολύ λιγότερο ελκυστικές. Το δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με τη σχέση ε, της Ενεργειακής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Ε, είναι αποτέλεσμα ε, συγκεκριμένης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής και ο στόχος είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση σε ε, αξιόπιστα, ε, φιλικά προς την ενέργεια και προς το περιβάλλον ε, σε φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις με σκοπό να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Και δεν υπάρχουν προγράμματα για την προώθηση των ορυκτών καυσίμων καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρική συμφώνησαν μέχρι το 2020 να έχουν τουλάχιστον 10.000 ΜΒ ε, ε, υδροελεκτρικής ενέργειας, 5.000 Β ε, αιωλικής ενέργειας και ένα σημαντικό όγκο επίσης παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια. Το τρίτο τμήμα Τη ερώτηση αφορούσε τους αναπτυξιακούς στόχου της χιλιετία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τους στόχου αυτούς ε, και ε, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρούμε ότι έχει, έχουν οι χώρες παρεκκλίνει από το στόχο τους και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό μέσω, για παράδειγμα, της δέσμευσης, της ταχείας δέσμευσης για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος το ερώτημα επίσης είχε να κάνει και με την, ε, το ρόλο με τις ε, ε, κυβερνητικές πρωτοβουλίες, πώς είναι δυνατόν δηλαδή η καλύτερη διακυβέρνηση να υπάρχει σε επίπεδο αφρικανικών, αφρικανικού θεσμικού πλαισίου. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα παρέμβασης και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε με σωστό τρόπο, ε, ώστε οι Αφρικανοί εταίροι μας να κάνουν μόνοι τους τις σωστή επιλογές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτζεντίνη. Ήταν μια πάρα πολύ διεξοδική απάντηση, δεν χρειάζεται να πω τίποτα κυρία Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Ναι, με συγχωρείτε. Για πίνγκ, θα έρθει λίγο αργότερα. Δεν μου έχουν πει κάτι από πλευράς Προεδρίας τουλάχιστον. Πάμε στο σημείο 5. Είναι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μήπως θα ήθελα να κάνω αυτές τις ανακοινώσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Όχι. Εντάξει. 7 Πρόκειται για την αποστολή την οποία έκανε η ε, εξεταστική αποστολή της Επιτροπής στο Πακιστάν υπό την ε, διεύθυνση του κυρίου Ντέβα ε, και ο κύριος Ντέβα θα μας παρουσιάσει αυτή την αποστολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είχα τη χαρά να ε, ηγηθώ μιας ε, πολύ ισχυρής επιτροπής σε τρεις μέρες και πήγαμε να δούμε ε, πώς έχουν χρησιμοποιηθεί οι πόροι που διαθέσαμε στο Πακιστάν ε, που ήταν η μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια που δόθηκε 150 εκατομμύρια για ε, να βοηθήσουμε την ανθρωπιστική κρίση που δημιούργησαν οι πλημμύρες από την αρχή διαπιστώσαμε στην αρχή των σχέσεών μας με το Πακιστάν ότι πρόκειται ε, για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή που διαπιστώσαμε 8 εκατομμύρια άτομα μετατοπίστηκαν και ε, υπήρχε μεγάλη φτώχεια μετακίνηση πληθυσμών έλλειψη υγειονομικών παροχών τροφίμων και ούτω καθεξής έπρεπε λοιπόν να πάμε να δούμε τι έγινε η ανθρωπιστική βοήθεια τα 150 εκατομμύρια και επιπλέον ε, ε, ε, ήταν ακόμη 153 εκατομμύρια και ποια άλλα ποσά τα οποία έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει το Πακιστάν στην αρχή πριν ξεκινήσει η ε, αποστολή αυτή υπήρχαν διάφορα θέματα σχετικά ε, με τον τρόπο με τον οποίο το Πακιστάν είχε διαχειριστεί την κρίση ε, ότι έπρεπε σε κάποιο σημείο να σταματήσει το ανθρωπιστικό θέμα και να προχωρήσουμε στην αναπτυξιακή φάση. Αλλά διαπιστώσαμε ότι οι συνομιλητές μας εις το Πακιστάν είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά και εδώ δεν, ε, ε, ε, δεν προσέχω τα λόγια μου είχαν βοηθήσει 1,5 εκατομμύριο άτομα τα οποία μπόρεσαν να επανέλθουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν να ευημερούν μέσα στους 9 μήνες μεταξύ της πλημμύρας και του χρόνου της επίσκεψής μας πράγμα το οποίο ήταν μια εξαιρετική επίδοση αν συγκρίνουμε με ε, τι έγινε ε, μετά το τσουνάμι που χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να μπορέσει κανείς να αποκαταστήσει το 1 τέταρτον αυτού του πληθυσμού σε χώρους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό λοιπόν το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι οι αρχές του Πακιστάν είχαν χρησιμοποιήσει το στρατό και ε, τίθεται θέμα στο Κοινοβούλιο εάν οι στρατιώτες πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν διαχειριστής ανθρωπιστικής κρίσης αλλά πρόκειτο για ένα εξαιρετικό παράδειγμα είχαν χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες που είχαν για να μεταφέρουν τους πολίτες με τον τεράστιο στρατό τον οποίο διαθέτουν με θαυμάσιο τρόπο και τώρα οι άνθρωποι αυτοί μας λέγουν ότι ε, δεν ε, πρέπει επίσης να αναφέρω ε, ότι δεν υπήρξε καμία επιδημία ούτε χόλερα ούτε καμία άλλη υπήρχε μια πολύ αποτελεσματική μηχανή για να μπορέσουν να αποκατασταθούν τα άτομα αυτά και όλοι όσοι ασχολούνται με ανθρωπιστική βοήθεια θα έπρεπε να ξανασκεφτούν να πρέπει να χρησιμοποιούμε τους στρατιωτικούς ε, για να σώσουμε ζωές διότι είδαμε ότι ε, υπήρξε ένα γεγονός το οποίο εμείς δεν είχαμε ε, προσέξει ε, και μετά από ένα χρόνο βλέπουμε ας πούμε στην Αϊτή το χάος και την καταστροφή και από την άλλη μεριά το Πακιστάν το οποίο μέσα σε εννέα μήνες προχώρησε τόσο πολύ. Για να μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε από την ανθρωπιστική φάση ή την αναπτυξιακή φάση χρειαζόμαστε ακόμη προσπάθειες αλλά πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγημεν. Όπως άλλωστε και οι συνάδελφοι βλέποντας πόσο αποτελεσματικά είχαν χειριστεί την κατάσταση. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις με τους πιο υψηλά ιστάμενους στο Πακιστάν. Συναντήσαμε τον ειδικό εκπρόσωπο από του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική πτυχή του, της βοηθείας του ΟΗΕ ε, και άλλους συμμετέχοντες οι οποίοι μας εδέχθηκαν ευγενέστατα ε, και αυτό ήταν δύο μέρες πριν το τέλος του Μπιν Λάντεν, ότως υπήν. Οπότε ε, ε, ήμουν ευτυχής όταν επανήλθα στο Λονδίνο αντί να παραμένω εκείνη την εποχή ή στα Πέριξ ε, στην Ινδία. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι είμαστε στο ξενοδοχείο Σιρένα 30 μίλια από εκεί που βρήκε το τέλος του ο Μπιν Λάντεν. Και τεκπλήξεως διαπιστώσαμε ε, τι είχε συμβεί. Συναντηθήκαμε λοιπόν με την κυρία Τίου Πακάλα που είναι η εκπρόσωπος ε, για τις ε, ανθρωπιστικές οργανώσεις και πρέπει να πούμε με πόσο αποτελεσματικό τρόπο ε, αποδόθηκε η ανθρωπιστική βοήθεια και πώς εφαρμόστηκαν τα διάφορα προγράμματα. Το πρόγραμμα ΕΚΟ πάντοτε είχε επενεθεί από τους ομολόγους μας για την αποτελεσματικότητά του. Υπήρξε και συνάντηση με έναν οικονομολόγο της ε, ε, Διεθνούς Τραπέζης σχετικά με τις επιπτώσεις των πλημμυρών στο Πακιστάν και όσοι από εσά έχετε επισκεφθεί τη χώρα αυτή ίσως γνωρίζετε ότι η ε, πρωτεύουσα και η υπόλοιπη χώρα είναι σε δύο διαφορετικούς οικονομικούς χώρους και αυτό είναι ε, ένα αστιάκι για την εικόνα του Πακιστάν. Δηλαδή η Ήπεθρος ε, ξεχωρίζει από την πρωτεύουσα και ε, είπαμε ότι υπήρχαν διάφορα προγράμματα για την ίδρυυση και την ε, υγεία μας έδωσαν βέβαια τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και ε, αστυνομικούς και περιπολικά με ανοιχτές τις ειρήνες οι οποίες ε, προπορευόντουσαν όπου πηγαίναμε αλλά εγώ στην πείρα που έχω από τον αναπτυξιακό χώρο είδα τους φτωχότερους ανθρώπους που έχω δει στη ζωή μου και αν φτωχοί είναι αυτοί που έχουν ένα δολάριο την ημέρα μπορώ να σας πω ότι εκεί ήταν στα 50 cents την ημέρα. Όλοι όμως μας εδέχθηκαν ευγενέστατα, μας ανέφεραν τα προβλήματά τους και τα προβλήματά τους είναι τα εξής. Δεν υπάρχει αποχέτευση στο χωριό και όλα τα, τα, απορρίμματα βρίσκονται σε μία τεράστια λίμνη γύρω από το χωριό. Και οι αρχές δεν είχαν τον τρόπο να δημιουργήσουν ένα αποχετευτικό σύστημα ή βόθρους ή άλλα πράγματα τα οποία θεωρούμε εμείς προφανή και θέματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθεί. Ε, υπήρχαν λοιπόν χιλιάδες μίνι ε, μήγες μέσα στα οποία συζητούσαμε πώς θα βελτιώσουμε το αποχετευτικό σύστημα στα διάφορα χωριά που είναι γύρω από την πρωτεύουσα. Έγινε μία συνάντηση με τον υποδιευθυντή της Επιτροπής Προγραμματισμού που εξέταζε τα μακροπρόθεσμα προγράμματα στο Πακιστάν γιατί είναι μια πολύ ασταθής χώρα και η αστάθεια αυτή και ο ευάλωτος χαρακτήρας εκφράζεται ε, μέσω των ε, περιορισμών. Δηλαδή βλέπουμε στα σύνορα με το Αφγανιστάν το πρόβλημα της ρομοκρατίας, την αστάθεια των Μπιν Λάντεν ε, και τους ακολούθιστους, τους Ταλιμπάν και πρόκειται για μια πυρνική δύναμη. Υπάρχει λοιπόν ένα μείγμα από πολύ περίπλοκες δομές δυνάμεις ε, και σκοτεινές κινήσεις όταν, ε, το οποίο διαπιστώσαμε όταν ε, μάθαμε ότι ο Μπιν Λάντινγκ διαβιούσε 30 μίλια από εκεί που ήμασταν και πώς δεν το γνώριζε το μισό Πακιστάν δεν το κατάλαβα. Όταν όμως συζητήσαμε τα προβλήματα αυτά με τις αρχές του Πακιστάν και ιδιαιτέρως με ε, τον ε, ε, Υπουργό Εξωτερικών Χίρνα Ραμπάνι Καρ, και συζητήσαμε τις ε, ε, μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις του να μπορέσει να έχει το Πακιστάν μία παραγωγή και που να εξαχθούν προς την Ευρωπαϊκή ή να βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις. Συζητήσαμε το GSP, το GSP Plus, το τι συνεπάγεται, που συνεπάγεται όχι μόνο το Πακιστάν να υπογράψει το CCPR, αλλά και να το εφαρμόσει στο πακιστανικό νομικό σύστημα. Το Κοινοβούλιο έχει κυρώσει τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί διεθνώς και τη συνθήκη κατά των βασανιστήριων και των ε, γυναικών ε, και ε, όλα αυτά τους είπαμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν. Είπαμε στον Πρωθυπουργό και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι πρέπει να κυρωθούν αυτές οι διεθνείς συνθήκες. Και ε, αυτοί σημείωσαν προσεκτικά όλες μας τις απόψεις και όλες μας τις απαιτήσει στον τομέα αυτό. Επίσης, αναφερθήκαμε στην ε, τροπολογία του άρθρου 18 της, του συντάγματος του Πακιστάν ε, το οποίο δεν, δια, ε, δεν αντιλαμβανόμαστε δηλαδή η μετακίνηση των εξουσιών από το Ισλαμαμπάντ στις επαρχίες είναι τεράστια και η τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείται με την αστυνομία, με τον ορυκτό πλούτο, με τα κίνηση και δεν υπάρχει καν μία ομοσπονδιακή δομή. Αυτό λοιπόν που με ανησυχεί είναι αν το κέντρο θα μπορέσει να συγκρατήσει τις παραμεθόριες επαρχίες στο σύστημα αυτό, το Βελουχιστάν, το Πουντζάμπ, και οι ε, βόρειες και ε, βορειοδυτικές περιοχές οι οποίες τώρα έχουν τοπική αυτοδιοίκηση με τρομερές εξουσίες κάτι το οποίο δεν είχαμε αντιληφθεί πριν από το ταξίδι μας δηλαδή δεν ξέραμε πόσο αποκεντρωμένη έχει καταστεί η διοίκηση του Πακιστάν και θέλαμε να εξετάσουμε αυτή την πτυχή, να δούμε πώς προχωράει αλλά και από πλευράς ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής προσπαθίας οι επαρχίες είναι αυτές οι οποίες θα ηγηθούν για να εφαρμοστούν τα μέτρα σε τοπικό επίπεδο και όχι από την πρωτεύουσα. Μετά όμως φύγαμε ξέσπασαν όλα τα δεινά ε, του φεκίστηκε ο, Μπιν Λάντεν δεν ξέρω ποια είναι η στάση εις το Πακιστάν ε, προς την Αμερική προς τη σταθερότητα ε, και εύχομαι η κυβέρνηση και το κράτος του Πακιστάν που έχουν ε, εδώ και ε, έξι χρόνια δημοκρατία μέχρι τώρα δυόμιση χρόνια και πολύ ήταν η πιο μακριά δημοκρατική περίοδος να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να τα βγάλουν πέρα. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβε για αυτά που μας είπατε, ήταν πολύ θετικά και τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής μια αντιπροσωπεία υψηλού κινέζικη για επαφέ με το εξωτερικό, αντιπρόεδρος κ. Λιγιαμπίνγκ, ε, παρατηρητέ της ε, συνάντησή μας. Ε, Καλώ ορίσατε. Το λόγο έχουν τα μέλη. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντέβα για την πολύ καλή του παρουσίαση, η οποία δείχνει βέβαια την αξία των ε, επί των αποστολών επιτόπου για την εξέταση μιας κατάστασης. Ε, επιτόπου μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών δράσεων από κοινού με άλλους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα ο ΙΕ. Και όπως είπε και ο κύριος Δίβα, και εμένα με ενδιαφέρει η συμμετοχή ε, των στρατιωτικών δυνάμεων όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανθρωπιστική δράση. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να τεθεί το θέμα του κατά πόσο ένας Αμερικανός στρα, ε, στρατιώτης πρέπει να, να ε, σώσει ένα παιδί από τη στέρηση, για παράδειγμα. Ε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να γίνει αυτό. Εντάξει, είναι σημαντικό βέβαια το ότι βοηθάμε κάποιον, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και γι' αυτό καταλαβαίνω, ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Ντέβα. Είναι μια καλή ε, ιστορία, ένα πολύ καλό παράδειγμα και είναι εξίσου καλό να βλέπουμε την ε, ιστορική εξέλιξη όπως επίσης και τις συνέπειές της στα ζητήματα που συζητούμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, σε, για όσους συμμετείχαν σε αυτήν ε, την αποστολή ήταν πάλι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και το λέω βλέποντας ε, το πρόγραμμά της είναι λοιπόν ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας φανταστικής δέσμευσης ε, πάρα πολλές ώρες δούλευαν τα μέλη της αποστολής και μάλιστα σπανίως ε, μας ε, επενούν γι' αυτό γιατί κανείς δεν θα το διαβάσει αυτό ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενδεχομένως να μην είναι πολύ σαφές πόσες ώρες περνάμε. Αρχίζουμε 8 η ώρα το πρωί και τελειώνουμε αργά το βράδυ. Θα ήθελα λοιπόν να πω προς τον κύριο Ντέβα ότι δεν μου φαίνεται καθόλου σύμπτωση το ότι μετά που φύγατε βρέθηκε ο Μπιν Λάντεν. Μάλιστα υπάρχουν οι φήμες ότι οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν ε, και μία επίσκεψη ε, στον ε, Μπιν Λάντεν και του είπανε «Τι θέλετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η η και είπαν εκείνοι «Όχι, όχι, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τέλος πάντων, πέρα από τα αστεία όμως, είναι καλό να βρίσκεται κανείς ε, σε χώρες ε, με τις οποίες έχουμε στρατηγικές σχέσεις, μακροχρόνιες σχέσεις, ακόμη και πριν από τέτοιου είδους συγκλονιστικά γεγονότα ή ακόμη και μετά, γιατί βλέπει κανείς πώς λειτουργεί μια χώρα και πριν αλλά και μετά από τέτοιου είδους συγκλονιστικά γεγονότα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε από ψυχολογικής απόψεως πώς εξελίσσεται μια τέτοια χώρα. Σε ξέρω πάρα πολύ καιρό, ε, Νάιρ, αλλά πραγματικά ο, ο ορισμός ε, που έδωσες ε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ περιγραφικός και θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ όλους όσους συμμετείχαν στην αποστολή γιατί ε, φαίνεται πάρα πολύ καλά στην έκθεση ε, πόσο πολύ δουλέψαμε για να μην ε, να ανακουφίσουμε ορισμένους ανθρώπους από την εξαθλίωση. Ο κύριος Γκέρενς. Ακούστε, από εδώ ξεκινάει η αφιβολία. Δεν ξέρω έτσι και αιτιατό ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κ. στο Πακιστάν και η, προ... η εξαφάνιση πρόορη του Μπεν Λάντεν. Τέλο πάντων μετά από αυτό. Να πω τη δεύτερη μου σκέψη. Χάρηκα που σας άκουσα να κάνετε τα σχόλια αυτά που μας ε, ρημούν αλλά και μας ανησυχούν. Το πρώτο γιατί όλες αυτές οι εργασίες μετά από τις πλημμύρες όλα αυτά προχωρούν πολύ καλά επειδή το Πακιστάν κυρίως ο στρατός έχουν πάρει στα χέρια στην κατάσταση, προχωρούν καλά τα πράγματα Όλα αυτά λοιπόν και τον Αύγουστο είχαμε εκδώσει ένα ανακοινωθέν ε, και εγώ ίδιος το έχω διαβάσει για το ότι χρειάζεται να δοθεί μια πολιτική κατεύθυνση στην κατάσταση και μια εξήγηση. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί το Πακιστάν είναι σημαντική χώρα αλλά και ιδιαίτερα ευάλωτη και όλα αυτά τα επενθυμίσατε στα όσα εισαγωγικά μας είπατε. Τώρα ε, τι γίνεται με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Πακιστάν, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, αν έχει εγκατασταθεί και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ακριβώς τι είναι, βλέπει ότι υπάρχει περισσότερη παρουσία στο Πακιστάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι οι Πακιστανοί και θα πρέπει να δούμε ακριβώς η εντύπωσή σας ε, πώς ε, την αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μια πραγματικότητα όλα αυτά που έκανε η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη αυτά τα έχουν αντιληφθεί οι Πακιστάνοι και μήπως με άνισο τρόπο μεταξύ τους. Ναι, σε αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσε να απαντήσει λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, η η... η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. I'm going to speak in θα μιλήσω ελληνικά. Σας δίνω όμως χρόνο για να βάλετε τα ακουστικά σας. Να Το ένα είναι ότι εκείνος που περιμένει την ανακουφιστική βοήθεια, την ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσει, αυτός που ζει με το μισό δολάριο την ημέρα, δεν κάνει διάκριση αν αυτό που του στέλνουμε είναι humanitarian or developmental aid Εκείνο θέλει να επιβιώσει και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Ήθελα και εγώ να πω στην αποστολή του στο Πακιστάν, αλλά δυστυχώ έμεινα έξω και χαίρομαι που ο κύριο Δέβα έχει επισημάνει τη σημασία τη συμμετοχή όλων των παραγόντων για την διάθεση, τη σωστή διάθεση τη ανθρωπιστική βοήθεια και του στρατού και οποιασδήποτε humanitarian task force και των εθελοντών και οποιονδήποτε. Επισημαίνω το γεγονό ότι το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη και συνεπώ εγώ θα επιμείνω στη θέση μου ότι οι χώρες που κατασκευάζουν πυρηνικά δεν πρέπει να περιμένουν αναπτυξιακή βοήθεια τη στιγμή που και οι ίδιες μπορούν να βοηθήσουν τον λαό τους να επιβιώσει. Τώρα, όσον αφορά τον Οσάμπα Μπιλάντεν, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να τελειώσω. Χωρίς να σημαίνει αυτό που θα πω ότι έχει λεχθεί κάτι το αντίθετο από τους προηγούμενους. Νομίζω ότι ήταν μια δολοφονία που δεν προάγει το σύστημα δικαίου στο οποίο κάποιοι από εμά πιστεύουν και θα έπρεπε να είχε γίνει μια διαφορετική, ένας διαφορετικός χειρισμός του, του ζητήματος. Δηλαδή με το να γίνεσαι χειρότερος από αυτόν που πας να τιμωρήσεις δεν δίνεις πολλές ελπίδες για το μέλλον. Και να σας θυμίσω την περίπτωση του Κάρατζιτς. Εδώ και τρία χρόνια τα μέσα τον καταδίκασαν και τον εκτέλεσαν δημόσια 20 φορές και όμως αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι γίνεται αυτή η δίκη. Εγώ ρώτησα την Επιτροπή πού βρίσκεται, είναι στις φυλακές, ζει, πέθανε, δεν ξέρω τέλος πάντων τι γίνεται με τον Καράτσιτς. Ευχαριστώ. Δεν σημαίνει βέβαια ότι υποστηρίζω την τρομοκρατία για όνομα του Θεού σε καμιά περίπτωση. Μη σκεφτεί κανεί να του δώσει διαστάσει που δεν υπάρχουν. Εγώ πιστεύω σε ένα σύστημα δικαιοσύνη που θα δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να υπερασπίζεται τον εαυτό του σωστά. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή θα πάρει το λόγο. Κυρία Κώστα, ξεκινώντας. Όχι. Πρόκειται για την ε, δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Πακιστάν. Αυτό αφορά η ερώτηση και αφορά επίσης την ορατότητα, της, ε, το πόσο γίνεται αισθητή η ε, δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε την ερώτηση πριν απαντήσω. Απλή ερώτηση. Προστιθέμενη αξία αυτής της νέας υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δηλαδή το αντιλαμβάνονται καλύτερα εδώ πολιτικά τουλάχιστον έτσι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνεται χάρη σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και τις αντιπροσωπείας ακριβώς που συμπράττει εκεί. Ναι. Μια απάντηση από την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων εκείνη αρμόδια. Και για τον κύριο Ντέβα η ερώτηση. Και από γυγλοπικής πλευράς τη φροντίσκευτη και σχετικά. Πριν από τον κύριο Μάριος, ε, θέλετε να απαντήσετε κύριε Ντέβα ή μετά. Ο κύριος Ντέβα. Ο κύριος Γκόρενς ε, πάλι με δυσκολεύει, με στριμώχνει με την ερώτησή του. Κοιτάξτε, πριν σας πω οτιδήποτε, θα ήθελα να καλωρίσω και εγώ τον Λι Πινγκ ε, που είναι ο αντιπρόεδρος ε, της ε, Ένωσης Φιλίας και τον Χι Φεν και τον κύριο Γκί η κυρία Ζαν Ρονίν, η οποία είναι πολύ παλιά μου φίλη από το Πεκίνο και ο Αντίν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η παρουσία της ΕΙΕΔ στο Ισλαμαπάντ δεν είναι τόσο προφανής. Προσπαθούν, αλλά ακόμη και στην πρεσβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μέσα στο διπλωματικό, στις διπλωματικές εγκαταστάσεις, είναι εκτός. Και υπάρχουν πάρα πολλές πρεσβείες, όπως για παράδειγμα των ΗΠΑ, Πολιτειών, της Κίνας, ε, της ε, ε, Μεγάλης Βρετανίας ε, που διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό και ιστορικό ρόλο στο πλαίσιο των διπλωματικών εγκαταστάσεων και των διπλωματικών κύκλων. Αλλά ο πρέσβης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ισλαμαμπάτ κάνει ό,τι μπορεί. Ήταν πραγματικά, μας βοήθησε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ διαθέσιμος, και κάνει πάρα πολύ δουλειά, μας βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε την αποστολή μας, ε, προσπάθησε να ε, διαπιστώσουμε ό,τι θέλαμε να διαπιστωθεί, οπότε θα ήθελα να του βάλω 10 για την προσπάθειά του. Ε, είναι γεγονός ότι η ΕΕΔ δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί τόσο καλά όσο θα έπρεπε ακόμη, ε, ενδεχομένως να είναι πολύ νωρίς, ξέρω εγώ τι να σας πω, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω πολιτικός. Ε, καταλαβαίνει ο κύριος Κέρενς την πολιτική μου άποψη για το θέμα αυτό, που άλλωστε αναφέρθηκε σε επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών της ε, ε, Μεγάλης Βρετανίας προς όλες τις πρεσβείες και τα προξενία σε όλο τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να σας κάνω περισσότερες, να σας πω περισσότερες εξηγήσεις αλλά ε, δεν ε, υπάρχει λόγος, ε, αναφερόταν, η ΕΕΒ να καθιστά εντελώς κενή κάθε προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι στο πλαίσιο των εξωτερικών μας επαφών. Τώρα κοιτάξτε για το ερώτημα, το ερώτημα το, το κατά πόσο είναι πυρηνική δύναμη και τι σημασία έχει αυτό. Κοιτάξτε, αν δεν σταθεροποιηθεί το Πακιστάν θα είναι ακόμη πιο επικίνδυνο το θέμα το, της πυρηνικής απειλής. Ε, αν το Πακιστάν ε, είναι ένα πλήρες μέλος της διεθνούς κοινότητας ε, και σταθερή χώρα, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να είναι ασταθές το Πακιστάν πάλι με πυρηνικά. Δηλαδή, να απαντήσω και στο ερώτημα έτσι της Ελληνίδας συναδέλφου μου. γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κύριος Γκέρενς ε, δεν θα χάσει την ευκαιρία ε, να σας ανταπαντήσει, όμως πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Μικρόφωνο παρακαλώ. Απλώς ε, ήθελα να κάνω μία προφανή δήλωση ότι η γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών της ε, Μεγάλης Βρετανίας ε, είναι μια προσωπική γνώμη που δεν εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εξωτερική, στην Επιτροπή Εξωτερικής Δράσης στον κύριο Μαριούς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε με τη σειρά μου θα ήθελα και εγώ εν ονόματι της Επιτροπής Εξωτερικής Δράσης να συγχαρώ τον ε, κύριο Ντέβα και τους συναδέλφους του για την πολύ επιτυχή ε, αποστολή. Αυτό που μου είπε ο κύριος Βίγκε Μάρκ ήταν ότι ήταν ιδιαίτερος ε, ευγνώμων ότι εποφεληθήκατε να θίξετε πολλά θέματα που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αρχές, ιδίως τις επιφυλάξεις ε, του Πακιστάν σχετικά με το ICCPR και το CAP και σας είμαστε πολύ ευγνώμονες γι' αυτό. Όσον αφορά το ρόλο της αντιπροσωπείας και του EES, στο Πακιστάν έχουμε βέβαια μία τελείως αποκεντρωμένη αντιπροσωπεία η οποία λειτουργεί καλά και είναι αποτελεσματική και τώρα θα αναλάβει την Προεδρία στο Ισλαμαμπάντ. Δηλαδή η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των συναντήσεων με τα κράτη-μέλη. Ο επικεφαλής έχει κάνει διαβήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ο συντονισμός της εργασίας είναι κάτι το οποίο έχει αυξηθεί. Όσον αφορά ε, ε, προγράμματα ε, θα πρέπει να υπάρχει μία κίνηση προς ε, την, ε, τον διπλωματικό θύλακο αλλά περιμένουμε ότι σε αυτό το διπλωματικό χώρο θα μπορέσουμε να έχουμε μία νέα εκπροσώπηση σύντομα. Η Πρόεδρος. Ακούστε, θα προχωρήσουμε στη συνάντηση για τις 65 τροπολογίες της έκθεσης του κ. Ντέβα για την ανέμωση των υποδομών φραγμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, την ίσχυση αυτών. Η διαχείριση για το νερό και για την επιβίωση των πληθυσμών εκεί και στην ε, περιοχή των παγετώνων στα Ιμαλάια επειδή αλλάζει το κλίμα και οι παγετώνες έχουν αβέβαιο μέλλον. Το λόγο έχει ο κύριος Ντέβα. Thank you, Madam Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. 67 είναι οι τροπολογίες ε, της συγκεκριμένης έκθεσης. Έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο στο Ευρωπαϊκό αυτό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι θα ψηφίσουμε αύριο ε, ως Επιτροπή και μετά να το στείλουμε στην Ολομέλεια. Γιατί είναι σημαντική η συγκεκριμένη έκθεση. Είναι σημαντική γιατί 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι και τα νοικοκυριά τους εξαρτώνται από την κατάσταση των συστημάτων υδάτων των Ιμαλαίων. Επειδή ε, λιώνουν ε, οι παγετώνες, ε, συμβαίνει το εξής τέσσερις φορές πιο γρήγορα ε, ε, λιώνουν οι παγετώνες αυτοί από ότι ε, του, των πόλων, από ότι των παγετώνων των πόλων. Ο λόγος λοιπόν που λιώνουν τόσο γρήγορα έχει ως αποτέλεσμα ότι πάρα πολλοί ποταμοί και στην Κίνα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή δεν θα έχουν καθόλου νερό. Και ο λόγος που δεν θα υπάρχει ε, νερό και ο λόγος που λιώνουν ε, οι παγετώνες, όπως είπα και προηγουμένως, ε, είναι το... From fires and cookers and wood. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει καθόλου να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει με αέρια τα οποία ε, μένουν πάνω στα Ιμαλάια με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία να απορροφάται περισσότερο, να λιώνουν πιο γρήγορα οι πάγοι και υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες παγετώνιες λίμνες, 300 ε, γύρω από τα Ιμαλάια, τα έχουμε φωτογραφίσει κιόλα, οι οποίες ε, μπορεί κατά ε, ανα χρονική στιγμή να πλημμυρίσουν τις γύρω, τις γύρω περιοχές, θα γίνει κάτι σαν έκρηξη δηλαδή, που θα δημιουργήσει μία πλημμύρα και είναι κάτι το οποίο βέβαια θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα και αυτό είναι ένα ε, πραγματικά ε, απίστευτο σενάριο, το οποίο όμως δεν είναι και τόσο απίθανο. Λοιπόν, ε, αν συμβεί κάτι τέτοιο και το αναφέρει αυτό και γι' αυτό η έκθεσή μου αναφέρει και την ίδρυση ενός οργανισμού του ΟΗΕ για το Μπουτάν, την Ινδία, το Πακιστάν, το ε, και άλλες χώρες για να σταματήσει, αυτέ, να σταματήσει το λιώσιμο των πάγων στα Ιμαλάια. Δεν κάνει τίποτε όμως ο ΟΗΕ και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να παρέμβει σε μια πολύ μακρινή περιοχή και να ε, δείξει στους φίλους και ε, γείτονες της ε, περιοχής ε, με 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, ότι αν δεν κάνουν τίποτα γρήγορα, πολλοί άνθρωποι θα πεινάσουν. Αυτό ουσιαστικά είναι ο στόχος της συγκεκριμένης έκθεσης, αλλά είχα προβλήματα στην δική μου επιτροπή, όταν μιλούσαμε δηλαδή για τις υποδομές, για τα φράγματα, δεν είναι μόνο το θέμα των φραγμάτων. Είναι είναι μια παγκόσμια κλιματική κρίση που υπάρχει, που έχει ξεκινήσει στα Ιμαλάια και κανένας δεν ε, την έχει λάβει υπόψη, ούτε καν ε, στο, στην ημερήσια διάταξη της Κοπενχάγης δεν ήταν. Πρέπει οπωσδήποτε να το προσέξουμε και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που οι Κινέζοι και Πακιστανοί φίλοι μου είναι εδώ. Μόνο ακόμη φίλοι από την Ινδία, το Πακιστάν και το Μπουτάν χρειάζεται ακόμα να συμμετέχουν για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε τι θα κάνουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντέβα. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Γκέρνης, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ο κύριος Κόγιετ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είχαμε πει ήδη στη συνάντηση του Μαρτίου. Για πρώτη φορά έχει ζητηθεί το θέμα αυτό και η Επιτροπή είχαν την υποχρέωση να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, να το εξετάσει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τη. Και σε σχέση με αυτό ακριβώ χαιρόμαστε που μπορούμε να σα εδώ στα μέλη σα ότι στα πλαίσια των δράσης μας για τις αλλαγές τις κλιματικές που είναι πρωτοβουλία φάρος μπορούμε να πούμε στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία σε θέματα μάχης κατά των κλιματικών αλλαγών. Για το 2011 το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει και μία δράση με το Μπουτάν και οι υπηρεσίες της αντιπροσωπείας μας ακριβώς διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση του Μπουτάν το πρόβλημα της στήξης των παγετώνων και αυτό το ε, σοβαρό πρόβλημα και με το ε, Υπουργείο Γεωργίας εξετάζεται και λιώνουν, ε, επαναλαμβάνω, οι πάγοι και εμείς εξετάζουμε πάντα το θέμα και έχουμε ένα νέο στόχο ο οποίος και προστέθηκε στην πρόταση για το όλο πρόγραμμα με μια οριζόντια προσήγγιση για να δούμε και τους κινδύνους ακριβώς λόγω της κλιματικής αλλαγής ε, και οτιδήποτε έχει σχέση και με κάθε κίνδυνο από την τήξη αυτή και θα συμπεριληφθεί λοιπόν όλα αυτά στην οριζόντια συζήτηση. Δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει πάντα με το πρόγραμμα δράσης ε, της ε, φορέα για αυτές τις αλλαγές. Για το 2012 θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ινστιτούτο Ισιμόντ με βάση το ΝΕΠΑΛ για θέματα όπως αυτό και με μια περιφερειακή περισσότερο προσέγγιση όπως ο κύριος Ντέβα το είπε πριν από λίγο γιατί το θέμα αυτό έχει διάσταση περιφερειακή βέβαια και επηρεάζει τα πράγματα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής αυτής. Επίσης τίθεται ένα πρόβλημα στην Λατινική Αμερική και ήρθαμε σε επαφή με συναδέλφους εκεί για να δούμε πώς μπορούμε να το λάβουμε και εκεί υπόψη μας, αν όχι στο σημερινό πρόγραμμα, τουλάχιστον ε, στην επόμενη φάση προγραμματισμού η οποία και θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Θα ήθελα να απαντήσω λέει ο κ η πρόεδρος. Ακούστε, ο κύριος Γκέρεντς που έχει ζητήσει τον λόγο και μετά ο κύριος Ντέβα. Euh, Ακούστε κάτι να σας εκμυστηρευτώ. Ότι δεν διαθέτω πείρα πάνω σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Ντέβα ε, το εξετάζει, είναι ιδιαίτερα λεπτό. Κάθε φορά που χρειαζόταν αυτές, αυτά τα μεγάλα έργα πάνω σε αυτό, όταν εξεταζόταν, ε, υπήρχε κάτι που ήταν πέρα από τον τεχνικό αυτό, καθ' αυτό χαρακτήρα του θέματος. Στα πλαίσια της έκθεσης πρωτοβουλίας ε, της συναδέλφου, θα πρέπει να κουμπίσουμε μια πληγή ουσιαστικά που τώρα ανοίγει και είναι η τήξη των παγετώνων στα Ιμαλάια και το θέμα το οποίο ασχολούμε θα είναι ακριβώς επίκαιρο και πρέπει να το εξετάσουμε όπως πρέπει. Θα πρέπει να δούμε σε αυτό το σχέδιο και τη διάρκεια του και χρειάζεται να ζυγίσουμε την το θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε και τις επιστημονικές απόψεις. Δεν ξέρω τώρα σε αυτή τη φάση αν γίνεται, αλλά είναι πρωτο... έκθεση πρωτοβουλίας. Εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε και καλό και χρήσιμο θα ήταν εμείς ε, τις ενέργειες αυτές που θα αναλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχουν και όσο γίνεται περισσότεροι εμπειρογνώμονες για να μην χάσουμε την ευκαιρία ξεκινήματος μιας καλής ιδέας ε, και χωρίς να έχουμε εξετάσει τις επιπτώσεις. Ε, η εξέταση αυτών είναι κάτι το πολύ σημαντικό και θα ήθελα να πω αυτά ακριβώς τα πράγματα στον κύριο Ντέβα. Βλέπετε πως περιφέρθηκα τη δεύτερη φορά σε αντίθεση με την πρώτη φορά. Κυρία μου. Ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή τον κύριο Ντέβα διότι είναι ένα πολύ βασικό θέμα και νομίζω επίσης ότι η χρυσή τομή βρίσκεται στη μέση ε, δηλαδή ε, υπάρχουν καταστάσεις όπου χρειάζονται φράγματα αλλά υπάρχουν και καταστάσεις όπου ε, δεν χρειάζονται και υπάρχουν οικολογικές σκοπιμότητες που μας υποκινούν να σκεφτούμε καλύτερα το θέμα του εάν χρειάζεται να κατασκευάζουμε φράγματα. Όχι απλά ναι, όχι ή κάτι τέτοιο, αλλά όπως είπε και ο κύριος Γκέρεντς, μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά πότε είναι σημαντικό διότι υπάρχουν άλλες περιοχές στον κόσμο όπου είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα δείτε σε ορισμένα σημεία ότι το θέμα της αυξήσεως και της ανόδου της στάθμης του νερού στο μέλλον θα μας απασχολήσει πολύ οπότε πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Η κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που άργησα τόσο πολύ και μπήκα από το αλλά είχα να παρουσιάσω μία έκθεση στην Επιτροπή Αλίας, οπότε έτρεξα. Ευχαριστώ τον κύριο Ντέβα για την έκθεσή του. Συμφωνούμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ε, ε, τις ε, ε, εκπομπές ε, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά στηρίζουμε τις προσπάθειες τις οποίες κάνει όσον αφορά την ε, επιτάχυνση της, ε, ε, των λιωμένων πάγων στα Ιμαλάγια δείχνει ότι οι περιοχές αυτές στην αρχή θα υποστούν πλημμύρες και μετά ξηρασία και η κατάσταση έχει χειροτερέψει σημαντικά διότι βλέπουμε ότι εάν λιώνουν η τήξη των πάγων δηλαδή στα Ιμαλάια μας υποδηλούν και μία άλλη ανάγκη να βελτιώσουμε τη διαχείριση του νερού για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε αυτές τις επιπτώσεις και τα μεγάλα προγράμματα φραγμάτων οδήγησαν σε μετατόπιση πολλών πληθυσμών και και ε, ε, σε ευάλωτα οικοσυστήματα όπως και κινδύνους ε, για τους πληθυσμούς που ζουν πιο χαμηλά από ό,τι τα φράγματα. Άρα υπάρχουν διάφορα επιχειρήματα για τα φράγματα, αλλά ένα μεγάλο φράγμα θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα από τα ειζήματα αργότερα και δεν ε, θα μπορέσει ε, να αντεπεξέλθει τόσο στις ανάγκες παραγωγής ηλεκτρισμού όσο και στην πρόληψη πλημμυρών όσο προβλέπουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας πολύ προσεκτικός προγραμματισμός προτού προχωρήσουμε. Η Επιτροπή Φραγμάτων μας τονίζει ότι πρέπει να ζητήσουμε τη συνένεση των εμπλεκομένων πληθυσμών κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες την υδροηλεκτρική παραγωγή, την αποθήκευση της ενεργείας και άλλους παράγοντες προτού προχωρήσουμε εις την κατασκευή των φραγμάτων. Έχουμε λοιπόν διατυπώσει πολλές τροπολογίες που προβλέπουν ακριβώς σε αυτούς τους στόχους και ελπίζουμε ότι ο εισηγητής θα συμφωνήσει μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι θα ήθελε να προσθέσει. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ο κ. Ντέβα έχει το λόγο, λοιπόν. Ευχαριστώ. Ας επανέλθουμε και ας εξετάσουμε το πρόβλημα αυτό λίγο παραπάνω. Διότι το πρόβλημα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μπορεί να το επιδεινώνει, αλλά ε, εάν μπει κανείς σε ένα ελικόπτερο και πάει 18.000 πόδια ψηλά, όπου δεν μπορεί καν να αναπνεύσει, μπορεί να δει ποιες είναι οι ατυχείς συσσωρεύσεις ε, ε, των υδάτων σε φυσικά φράγματα, όχι ε, κατασκευασμένα από τους ανθρώπους. Και εκεί έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ νερό. Γιατί συσσωρεύεται το νερό, το νερό συσσωρεύεται διότι υπάρχει υλοτομία ιδίως στην ε, Ινδία και στο Πακιστάν και τα δέντρα αυτά α, καίγονται σε σόμπες, ε, ξυλόσομπες που δημιουργούν την, καπνιά που ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, δημιουργεί αυτό το σύννεφο και επιταχύνει την τήξη των πάγων. Οπότε υπάρχει μία αλυσίδα. Κόβουμε τα δάση και με τα ξύλα δημιουργούμε την ε, ε, καπνιά ε, η οποία εμποδίζει την καθαρή ατμόσφαιρα ε, είναι δηλαδή μη ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί από τις χώρες που είναι γύρω από τα Ιμαλάια να σταματήσει η κοπή των δένδρων και η ε, καύση του ξύλου. Γι' αυτό και το νερό λιώνει τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι στον ε, ε, Βόρειο Πόλο. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτές τις θυματολογικέ αλλαγές τις οποίες θέλουμε, τότε ε, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα δέντρα από το δάσος ε, για να μειωθεί και η μαύρη καπνιά ε, μπορούμε να δούμε ε, τις ε, λίμνες αυτές. Έχω 300 φωτογραφίες από 300, φυσικούς, ε, από 300 φυσικές λίμνες. Είναι λοιπόν κάτι όπου η Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπουτάν και η Κίνα πρέπει να συναντηθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό. Διαφορετικά θα ξεφύγουν τελείως τα ποτάμια αυτά, θα αποξηρανθούν, τα μεγαλύτερα ποτάμια της Κίνας θα αποξηρανθούν όπως και της Ινδίας και αυτό είναι μέρος του τεράστιου παγκόσμιου προβλήματος το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τις τεχνικές τροπολογίες και το γραφείο μου είναι πολύ ευγνώμων για τις τροπολογίες και με τα θα δεχτώ ορισμένε από αυτές. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Ε, η ψηφοφορία αύριο 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί, θα διεξαχθεί. Εντάξει. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο, το 8, για τα τρόφιμα. Και έχει στηθεί ένα έγγραφο της 25 Ιανουαρίου και για την έκθεση αυτή το λόγο έχει η κυρία Τσίμερ. Έχει το λόγο η κυρία Τσίμερ, η συγγήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτή την έκθεση ε, στην Επιτροπή γιατί με βοήθησε να μάθω πολλά πράγματα από το γεγονός και μόνο ότι και στη δημόσια γνώμη αλλά και πέραν από την Ευρώπη το θέμα της διατροφικής ασφάλειας και των τροφίμων έχει ε, προσελκύσει μεγάλη προσοχή τους τελευταίους μήνες και το ενδιαφέρον για την έκθεση αυτή. Ξεπερνά τα πλαίσια της Επιτροπής μας αλλά και τα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ουσιαστικά επηρεάζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κατάρτιση ε, των μη κυβερνητικών ε, ε, των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Βλέπουμε δηλαδή ότι πρέπει να βρούμε πιο συγκεκριμένα σημεία στα οποία πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα και που πρέπει να επέμβουμε. Αλλά στα πλαίσια αυτά μας έχουν προσεγγίσει διάφορες οργανώσεις όπως ο ΙΕΙ, η ΟΥΚΤΑ, η UNIDO, η ΦΑΟ, προγράμματα της ε, ε, προστασίας και πρόθεσης της διατροφικής ασφάλειας πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδουν μεγάλη σημασία στον τομέα αυτό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Βαλερή Ραμέ η οποία με στήριξε τουλάχιστον εμένα προσωπικά εκ μέρους ε, από πλευράς της γραμματείας για, κατά την κατάρτιση αυτού του σχεδίου και να ευχαριστήσω επίσης και τους χειώδεις οσηγητές οι οποίοι από την αρχή προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν. Λυπάμαι ότι δεν μπορέσαμε ε, μέχρι τον Ιούνιο να διοργανώσουμε αυτήν την ακρόαση που είχαμε προβλέψει και η οποία πρέπει να αναβληθεί μέχρι την παρέλευση του καλοκαιριού και ελπίζω ότι θα μας επιτρέψει να γίνει η ακρόαση αυτή με τις διάφορες διασυνδέσεις της για να επιστήσουμε την προσοχή ε, της κοινή γνώμης από αυτού του θέματος και για να προωθηθούν ορισμένα προγράμματα. Εν τω μεταξύ στο σχέδιο αυτό ουσιαστικά στηρίζομαι στις δύο ανακοινώσεις τις οποίες δημοσίευσε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μία ανακοίνωση για την στήριξη των υποανάπτυξη χωρών για την βελτίωση της διατροφικής ασφάλειας και για την προώθηση του τομέα της διατροφής. Βλέπουμε όμως ότι το πλαίσιο αυτό δεν επαρκεί καν και ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποια επεξεργασία για να διευρυνθεί η ποικιλία των θεμάτων και επ' αυτού έχω τονίσει ότι στα πλαίσια αυτής, της, αυτού του σχεδίου ο εκθέσεως θέλω να σας ενθαρρύνω κατά τρόπον ώστε η διατροφή ε, δεν υπάρχει ακριβής όρος στα γερμανικά που να ε, περιγράφει το πρόβλημα αλλά ε, το ασυστατικά της διατροφής, την ποιότητα της διατροφής, η καλή διατροφή πρέπει να τύχει προσοχής και γι' αυτό ελπίζω ότι μέχρι την επόμενη περίοδο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια σχετική ανακοίνωση κατά τρόπον ώστε να εμβαθύνουμε τη συζήτηση για τη γεωργική πολιτική, για την ενεργειακή στρατηγική και για την κατάρτιση των θέσεων τις οποίες θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο G20 και σε όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει για να καταδείξουμε σε εστιασμένες και συγκεκριμένες κινήσεις ε, των ε, κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων για να μπορέσει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό διότι όσον αφορά ε, την διατροφική κρίση έχουμε ξεπεράσει την έκταση της κρίσης του 2008. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εφέτος, αλλά σύμφωνα με την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων, νομίζω ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου και πρέπει να αποδοθεί μεγάλη σημασία και προσπαθώ άλλωστε στην έκθεση να θέσω ε, το ερώτημα που αναφέρεται σε την διασύνδεση του δικαίου με τα τρόφιμα ξέρω ότι είναι ένα φιλεγόμενο θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως και στην Επιτροπή μας ε, πιστεύω ότι και στον τομέα των τροφίμων πρέπει να υπάρχει κυριαρχία και είναι απαραίτητος ε, ε, βάσιμο να γνωρίζει κανείς τι παράγεται σε τοπικό επίπεδο, τι χρειάζονται οι διάφοροι πληθυσμοί και νομίζω ότι εδώ καλό θα ήταν να μπορέσουμε να υποκινήσουμε τους παραγωγούς και την τοπική αυτοδιοίκηση να εμπλακούν πολύ πιο ενεργά από ό,τι συνέβη στο παρελθόν. Αλλά αυτό το οποίο ε, ε, μου προκάλεσε ορισμένες επιφυλάξεις είναι ορισμένες αξιολογήσεις οι οποίες επιβεβαιώτηθηκαν σε ορισμένα θέμα και που θα ήθελα να τονίσω εδώ. για να μπορέσουμε να επιτύχουμε στον αγώνα για την ε, φτώχεια και την πείνα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την κατάρτιση μίας, μία, μίας τροποποιημένης αναπτυξιακής πολιτικής. Αν η πείνα παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν το ποσοστό των επενδύσεων εις ε, την ε, γεωργία να έχει μειωθεί σημαντικά κατά την τελευταία τριακονταετία. Χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται νέες προτεραιότητες, πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο και επίγον. Όσο αναφορά το έγγραφο εργασίας, το οποίο ε, καταρτίστηκε για την ε, Επιτροπή. Ορισμένοι σκιώδεις εισηγητές ε, αλλά ε, και συντονιστές τονίζουν το θέμα της κερδοσκοπίας στις πρώτες ύλε και στα τρόφιμα και θεωρούμε ότι πρέπει να τονίσουμε ότι η πρωτοβουλία της Γαλλικής Προεδρίας στο G8 πρέπει να στηριχτεί. Είναι ένα θέμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μία πιο δεσμευμένη αντιμετώπιση ε, και ε, πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική κερδοσκοπία στα τρόφιμα, στις πρώτες ύλες. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και όταν δεν πρόκειται για πραγματικές ε, προθεσμιακές πράξεις μιλάμε ε, για ε, γεωργικά προϊόντα τα οποία πρέπει να διατίθενται εγκαίρως στην αγορά και άρα εδώ πρέπει να περιοριστεί η κερδοσκοπία και αυτό είναι μια κοινή μας ευθύνη την οποία πρέπει να αναλάβουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θεωρούσα ως σημαντικά και ήθελα να τα συζητήσουμε και σας αναφέρω ότι ε, στην Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε την ε, σημασία των μικρών ε, γεωργών και αγροτών και εγώ έχω παραπέμψει επανειλημμένος έχω επισημάνει με συγχωρείτε επανειλημμένος ότι ε, το 80% των ατόμων στις ανάπτυξης χώρες εργάζονται στη Γεωργία και το 90% εξ αυτών δεν μπορεί να αυτοσυντηρηθεί ικανοποιητικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ορισμένες ε, αλλαγές στην παγκόσμιο πολιτική και γι' αυτό ε, εγώ παρουσιάζω μία μία θέση την οποία θεωρώ βασική ότι δηλαδή η συνένεση της Ουάσιγκτον οδήγησε στο ότι η απέτηση μεγάλης απελευθέρωσης και μείωσης των δασμών πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει σταθεροποιήσει την διατροφική ασφάλεια ανά τον κόσμο αλλά μάλλον έχει προωθήσει την αντίστροφη εξέλιξη. Σαν Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε υπεύθυνοι και οι στόχοι μας στην ενεργειακή στρατηγική και πολιτική πρέπει να αποβλέπουν σε μια βιώσιμη ε, πολιτική ε, και δεν πρέπει μεγάλες εκτάσεις χωραφιών να διατεθούν ε, για να καλλιεργούνται πρώτες ύλες ενεργείας που αναπτύσσονται γρήγορα και Πέραν αυτού, πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει γιατί συνάντησα μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον μία ανακοίνωση η οποία αναφέρεται εις την πολιτική της υπαίθρου που δεν γνώριζαν οι περισσότεροι και σχετικά με το πλαίσιο αυτό για μια πολιτική της υπαίθρου διαπιστώσαμε ότι πάρα πολλές χώρες ακολουθούν το δικό τους δρόμο αντί να κινούνται ε, συλλογικά οι χώρες και να είναι πιο συνειδητοποιημένες. Δεν πρέπει δηλαδή πλέον κανείς εδώ να εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα αλλά να υπάρξει ε, μία εξέλιξη που θα είναι διαφορετική από αυτή που οδήγησε ή στην οικονομική κρίση, στην πετρελαϊκή κρίση, στη διατροφική κρίση όπου βλέπουμε ότι ε, χώρες αγοράζουν ε, εκτάσεις τις οποίες έχουν αφαιρέσει από τους παραγωγούς ε, έτσι προσπαθώ να διαμορφώσω την έκθεση αυτή. Υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να θίξουμε, αλλά επειδή η έκθεση αυτή πρέπει να είναι σύντομη, δεν μπορεί να τα καλύψει όλα και θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια αυτά, μέσω των τροπολογιών, να εμπλουτίνουμε το κείμενο και απλώς σας αναφέρω το πρόβλημα των αποβλήτων των τροφίμων που είναι ένα βασικό μέτρο προστασίας από την κακή διατροφή και την υποσύτηση και πρέπει να κοιτάξουμε με την δημοκρατική εξέλιξη τι ανάγκες διαμορφώνονται ε, για την διατροφή του πληθυσμού και πώς θα επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό πολιτικά. Ε, ε, προτάσεις ε, περιορίστηκα στις προσωπικές μου απόψεις διότι πιστεύω ότι σε ορισμένες χώρες συζητείται μία λανθασμένη ε, στρατηγική όπου οι χώρες δεν λαμβάνουν υπόψη την αύξηση του πληθυσμού ε, και δεν αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να τροφοδοτήσουν περιοχές της γης όπου ο πληθυσμός αυξάνεται ταχαίως. Και το λέω αυτό ε, γιατί η άποψη αυτή δεν πρέπει να υπερισχύσει. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με την παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τσίμερ για αυτή την τόσο καλή έκθεση. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατήρησεις. Σίγουρα αυτή η επιστική ασφάλεια είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Θα πρέπει να είναι στο πρώτο πλάνο των θεμάτων που εξετάζουμε. Σας κατανοώ όταν λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τη γεωργία στα πλαίσια της βοήθειας για την ανάπτυξη Δηλαδή, δημοσιομικός μηχανισμός καινοτόμος όπως ένας φόρος συναλλαγών ε, οικονομικών ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συμπληρωματικά κονδύλια και να βοηθήσουμε τους, ε, στους ευαίσθητες χώρες, τους περισσότερο ευάλωτους και για ένα δισεκατομμύρια ευρώ δύσκολα είναι να δούμε όλα αυτά πώς επηρεάζουν τα πράγματα για την πείνα και το αιτιοαιτιατό και πολλές φορές είδαμε αυτά πρώτην Επιτροπή ότι δεν υπήρχε πρόσβαση τις μικρές μεσαίες εκμεταλλεύσεις οικογενειακού χαρακτήρα, κυρίως από γυναίκες και από φτωχό πληθυσμό που, κρύ, που θίγει αυτή η κρίση και επίσης τις εξαγωγές μετά το 2013 στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που εξάγονται στον ΠΟΕ και να δούμε την ε, νομική δυνατότητα επιστροφής στις εξαγωγές σε περίπτωση δινής κρίσης όπως το 2009 για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και έτσι συγκυριακά να ελαφρύνουμε τους ε, παθόντες εισαγωγικά και επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερα την ε, Ανάπτυξη της βοήθειας ανθρωπιστικής και όλα αυτά με τις σχέσεις, μια αποκατάσταση, μια ανάπτυξη, όλα αυτά τα μέτρα και γι' αυτό προτείνω και σχετικές τροπολογίες. Ο κ. Μπέρμαν θα συνεχίσει. Έχετε το λόγο κύριε Μπέρμαν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι εξαιρετική και δείχνει πόσο έχει αλλάξει το πλαίσιο σε σχέση με την ανάπτυξη της υπαίθρου και με την ε, αγροτική, τη γεωργική πολιτική και τη σχέση της με την, με την αναπτυξιακή ε, βοήθεια. Όταν μειώθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό λοιπόν η σχέση μεταξύ αυτών των τομέων ε, Είναι κρίμα βέβαια που πλέον έχει αντιστραφεί η τάση. Είναι, είναι καλό που έχει αντισταθεί, αντιστραφεί η τάση δεδομένου ότι υπήρξαν πολλές επισητιστικές κρίσεις ε, οι οποίες ε, σήμεραν ότι κάτι τέτοιο ήταν επιτακτικό. Είναι λοιπόν καλό που άλλαξε αυτή η τάση. Μία ακόμα παρατήρηση. Η Πατήσια Τόια δεν μπορεί να είναι εδώ σκιώδη συγχύτρια για τους ε, σοσιαλδημοκράτες και δεν μπορεί να παρουσιάσει εκείνη τη δική της άποψη για την εξαιρετική έκθεση της Γκαμπριέλ Τσίμερ. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα ακόμη. Νομίζω έχετε απολύτως δίκιο όταν ε, τονίζεται την ε, ανάγκη αντιμετώπισης της κερδοσκοπίας ε, στα αγαθά και την ανάγκη ρύθμισης των αγορών όταν υπάρχουν παράγωγα ε, επί των ε, προϊόντων, επί των τροφίμων. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της αρπαγής της γης σε πολλές περιοχές. Είναι σημαντικό να μεταρρυθμιστεί η ΚΑΠ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζει πλέον ε, την γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο απεσιόδοξος προς αυτό γιατί δεν, ε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές το πλαίσιο του, του πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για αλλαγή, για την ανάγκη προσαρμογής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ε, στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Μόνο για τα συμφέροντα μιλάμε και η ιδέα ότι μπορεί κάποτε στο μέλλον ε, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις να καταργηθούν ε, απορρίφθηκε από σχεδόν όλους και πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το θέμα είναι ντροπή, δεν θα έπρεπε να υφίσταται καθόλου. Έχουν εξαφανιστεί από 10 δισεκατομμύρια σε 3 εκατομμύρια σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να εξαλειφθούν εντελώς. Κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να πω, Γκαμπριέλα, στο άρθρο 3... Όταν λες ότι κάνεις έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναπτυξιακό πρόγραμμα και να αυξήσει ε, τα προγράμματά της υπό τη τα προγράμματα ε, υπό τη διεθνή ηγεσία. Εγώ νομίζω ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου κυρίως ε, πρέπει να ενισχυθεί. Ήμουν στην ε, βορειοανατολική Κένια της, ε, προα... της προάλλες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ξηρασία, ε, ε, μη γόνιμες περιοχές και υπάρχουν άνθρωποι απεγνωσμένοι που ψάχνουν νερό μέσα στην άμμο. Είναι σαφές ότι αυτό που χρειάζεται εκεί για να μπορέσει κανείς να επιβιώσει ως, γεω... ως γεωργός, ε, ως ένας άνθρωπος που έχει ας πούμε μερικές ε, γίδες απλώς ε, χρειάζονται και σχολεία, χρειάζεται κάποια ε, υγειονομική περίθελψη για τους ανθρώπους, χρειάζεται μια ολόκληρη υποδομή που δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης ανάπτυξης της υπαίθρου. Δεν είμαστε λοιπόν υπέρ της γεωργίας, είμαστε υπέρ της ανάπτυξης υπαίθρου γενικότερα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, επαναλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Ακόμη αναφέρεται και στο θέμα τη ε, ε, επισυτιστικής κυριαρχίας ε, που είναι κάπως ταμπού σε γεωργικές συζητήσει. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ ο κύριο Γκέρεν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τσίμερ ε, αξίζει γιατί συνέταξε μια πολύ σημαντική έκθεση με έξυπνη σύνταξη. Συζήτησα μαζί της ε, κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς που δεν φύστηκε προσπαθειών ακριβώς πάνω στο θέμα αυτό. Οι παρατηρήσεις ε, δεν αφορούν την έκθεση αυτή, αλλά το θέμα της η στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο πρόβλημα που έθιξε η κυρία Τσίμερ ήταν ε, μια ιδιαίτερη αντίδραση. Θυμάστε ότι η διεθνής κοινότητα να είχε ασχοληθεί με αυτό πριν από πέντε χρόνια όταν ε, ε, το είχαμε ξεκινήσει για πολλά πολλά χρόνια Υπήρξε σιωπή και ξεκίνησαν τότε να μιλάνε για τη γεωργία, χωρίς όμως να υπάρχει μια κατάλληλη συνοχή στην όλη συζήτηση. Να μιλήσω για την έλλειψη συνοχής και για τις υπερβολές επίσης. Αντίθετα με αυτά που είπε συνάδελφος, συμφωνώ βέβαια, ότι δεν μας φτάνει να αυτομαστιγωνόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο Αυτές οι επιδοτήσεις στις εξαγωγές ε, έχει υπερτιμηθεί αυτό και τον αγνώρισε όταν το πρόβλημα το 30 μέσω αυτών των, της βοήθειας και παραμένει το θέμα ως έχει και λείπει μια κάποια συνοχή. Εδώ και αρκετά χρόνια είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο και πάντα οι ίδιες συζητήσεις επαναλαμβάνονται παρόλο που τα στοιχεία έχουν αλλάξει θα πρέπει εμείς ε, να κοιτάξουμε ακριβώς σε αυτούς μας, ε, να δούμε τι έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι. Και επίσης ε, είχε τη σοφία να δείξει τα κύρια σημεία της στρατηγικής για την προσπάθεια εξέβρεσης μιας λύσης στο πρόβλημα το γενικό της, του και επίσης ε, εδώ δεν υπάρχει μόνο οικονομική διάσταση και μόνο για τρόφιμο. Εδώ όλο το σύνολο ισχύει και θα πρέπει να δούμε και τις αδυναμίες ε, ε, να αυτού του συστήματος. Ε, μας έρθει να βάλαμε τις φωνές όταν δούμε αυτά τα πράγματα. Η ΦΑΟ έχει μελέτη ακριβώς επιπτώσεων σχετικά με την κατάσταση εδώ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ και πολλά χρόνια ε, ψάχνω να βρω μια μελέτη που να αξίζει το όνομά της σχετικά με τη ΦΑΟ που ασχολείται ακριβώς κυρίως αυτή πρώτη με αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να πληρώσουμε το κενό αυτό, να το καλύψουμε και ακόμα κάτι. Πρώτα απ' όλα, κυρίως βλέπουμε μια αδυναμία των αναψωμένων χωρών να μπορέσουν τα ίδια να οργανωθούν όπως πρέπει και να μας πούν τι δεν πάει καλά. Το ιδιαίτερα δραματικό στο όλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η αδυναμία για να προσφερθεί μια συντονισμένη απάντηση σε αυτά τα προβλήματα στερεί έτσι από τις αναπτυσσόμενες χώρες από το βασικό δικαίωμα, το θεμελιώδες που είναι η διατροφή, και αυτό βλέπουμε διάφορες εμπορικές βιομηχανικές ε, εταιρείες και τα κράτη-μέλη αντιποκαθιστούν τους υπόλοιπους. Ε, σκάνδαλο είναι. Γιατί, όχι γιατί αγοράζουν γη, αλλά γιατί τα χώρες αυτές δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα επιλογής. Δηλαδή να μπορέσουν να έχουν ε, τις απαραίτητες πηγές, τις απαραίτητες πόρους για να προχωρήσουν την παραγωγή των τροφίμων που χρειάζονται. Εδώ λοιπόν Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω για μία δήλωση του Μπιλ Κλίντον στην Αμερικανική Γερουσία μετά από το σεισμό της Αιτίας, ο οποίος εξομολογήθηκε ακριβώς ότι ναι, ήταν υπεύθυνος επειδή δεν μπορούσε η ΑΕΤ σήμερα να παράξει αρκετά προϊόντα διατροφής. Όσοι γνωρίζουν τη ιστορία της ΑΕΤ θα δουν μέχρι το σημείο αυτή η δυνατότητα γεωρικής παραγωγής μειώθηκε αυτά τα τελευταία 50 χρόνια. Πρόκειται για σκάνδαλο, αληθινό σκάνδαλο και είχε το θάρρος να το εξομολογηθεί αυτό ο να πει ήταν φταίξιμό του επίσης και ήταν συνυπεύθυνος επαναλαμβάνομαι για την κατάσταση αυτή και είπε ότι είδε τα θέματα τα εμπορικά όσα έχουν σχέση ανάμεσα στις βιομηχανικές χώρες και στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς τα θεμελιώδη δικαιώματα του καθένα όπως αυτή, το δικαίωμα του να τραφεί και με μια παράφραση των όσων είπα η κυρία Τσίμερ, ε, μάλλον τα χρησιμοποίησε όμως αφού τα άλλαξε κάπως ε, και είναι προς τιμή της. Ε, εντάξει, θα πρέπει να είναι σχεδόν μόνιμη η συγγήτρια για τα θέματα αυτά Υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν στην επιτυχία και άλλες δρόμοι στην αποτυχία. Η Ζιμπάμπουε μας έδειξε δρόμο τι δεν πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το μονοπόλιο μερικών που έχουν τη γη. Γιατί αν την λάθος θέση κανείς υιοθετήσει τότε αφισβητούνται τα πάντα. Αλλά μέσα σε, όπως συνέβη στη Ζιμπάμπου, αλλά στα πάντα και στο τίποτα θα πρέπει να είμαστε εμείς για να υποβάλουμε έξυπνες προτάσεις. Και πάλι αυτό είναι παραπονό μου εδώ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να δούμε πώς μπορούν να συνδυαστούν ε, τα ε, να αρθρώσουν λόγο και να πούν τις προτάσεις τους αυτά να βγάλουν κραυγή απόγνωσης να πούν ότι εδώ μας τερείται το θεμελιώδες δικαίωμά μας και όποιος δεν έχει δυνατότητες επιλογής τότε τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά η έκθεση της κυρίας Τσίμερ είναι άριστη βάση κατά την άποψή μου για να συνεχίσουμε έτσι να το σκεφτόμαστε, να το αναλύουμε. Είναι τρομερά σημαντικό το θέμα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να την ευχαριστήσω άξονόματος της ομάδας μου. Ευχαριστώ όλοι πρόεδρος και τώρα ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ χαιρετίζω την έκθεση αυτή και ευχαριστώ τη συνάδελφο Τσίμερ ε, για την εισαγωγή και τα σχόλια που έκανε. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με το πνεύμα της έκθεσης. Εγώ ήμουν εισηγητής ε, για την νομοθεσία για την έκτακτη επιστηστική βοήθεια και πολλοί κόσμος ε, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα σε διάφορες χώρες γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν αρκετά τρόφιμα. όταν ε, ερχόμουν σε επαφή με το Συμβούλιο Υπουργών έλεγαν ε, ότι 20 στους 27 δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτό που ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα έκτακτο κονδύλι 20 εκατομμυρίων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, τελικά τα καταφέραμε βέβαια γιατί απειλήσαμε να το πάρουμε από το πλεόνασμα της ε, γεωργικής πολιτικής όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε ολόκληρο το δισεκατομμύριο μέσα σε μία χρονιά. Τα καταφέραμε αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Αν είχαμε αυτήν την στάση από την αρχή, δηλαδή ο κόσμος πεινάει, δεν υπάρχουν τρόφιμα, ε, είχαμε αυτή τη στάση από την αρχή, θα είχαμε περισσότερο χρόνο νομίζω να σκεφτούμε και να ε, προετοιμαστούμε. Εγώ πιστεύω στις, ε, στην ελεύθερη αγορά. Νομίζω όμως ότι μερικές φορές όταν μιλάμε για ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για πραγματικά ελεύθερες αγορές, μιλάμε για ελεύθερα μέσα ενημέρωσης ε, που πολλές φορές δημοσιογράφοι κάνουν αυτό που θέλουν τα αφεντικά τους γιατί εκείνοι, εκείνα τους πληρώνουν. Και νομίζω ότι και στι αγορές υπάρχουν άνθρωποι που χειραγωγούν τις αγορές αυτές και νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της κερδοσκοπίας για τα ε, τρόφιμα και ο συνάδελφος ε, καλώ έθεσε το θέμα αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν ενδιαφέρονται για τις συνέπειε εφόσον εκείνοι θα κερδίσουν. Όταν βλέπουμε λοιπόν ολόκληρη τη διοντολογία του πώ λειτουργούν τα πράγματα, ε, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί σωστά θέτει το θέμα η κυρία Τσίμερ ε, ε, των διατροφικών στοιχείων, των θρεπτικών στοιχείων. Υπάρχει ένα πρόβλημα παχυσαρκίας στις ε, ανεπτυγμένες χώρες, γιατί οι άνθρωποι τρώνε λάθος φαγητό ή εν πάση περιπτώσει το φαγητό που είναι διαθέσιμο έχει πάρα πολλά λιπαρά, δεν ξέρω ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν δείτε κανείς πόσοι πεθαίνουν από μη μεταδοτικές ασθένειες, για παράδειγμα ο Bill Gates πριν από μερικές εβδομάδες είχε πει κάποια πράγματα που με έκαναν να αλλάξω την άποψή μου για τις ε, μη μεταδοτικέ ασθένειες. Πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι και ειδικώ γυναίκες, κυρίως γυναίκες, πεθαίνουν από ε, ε, ανακοπή καρδιάς που δεν είναι μια μεταδοτική ασθένεια και νομίζω ότι η διατροφή στο θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκέρεντς ήταν πραγματικά ε, σοκαριστικό να βλέπουμε τι συνέβη στην Αφρική αλλά κατά τη διάρκεια της ε, περίοδου που εγώ ήμουν εισηγητής για το θέμα που ανέφερα προηγουμένως της επίγουσας επιστητικής βοήθειας υπόθηκε το εξή. Έχουμε ένα πλεόνασμα. Μπορούμε να, να ταΐσουμε το Βιετνάμ ε, και την Βυρμανία και η εντύπωσή μου ήταν ότι μπορούσαμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούμε με περιφερειακούς οργανισμούς, ε, ε, με, με χώρες σε κάποιο φόρματ ομίλων, εν πάση περιπτώσει, και να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε μαζί τους για να βοηθήσουμε τις ε, περιοχές αυτές. Αναρωτηθήκαμε όμως γιατί Μπορεί η Ιρλανδία ας πούμε, να εξάγει τρόφιμα όταν χώρες... Ε, ε, ε γιατί, οι γειτονικέ χώρες ας πούμε ε, αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα επισητιστικά προβλήματα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από μόνο του. Αν κάποιοι έχουν μία γη να καλλιεργήσουν και έχουν τη δυνατότητα να το καλλιεργήσουν, θα μεταχειριστούν την, ε, την γη αυτή με διαφορετικό τρόπο, θα προσπαθήσουν να ε, παράγουν επαρκή τρόφιμα για, τον, για τις οικογένειές τους. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να είναι έξυπνοι ε, ε, γεωκτήμονες για να το πω έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε αυτό το θέμα και είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει συνεχώ ενδεχομένω να το παρακολουθούμε. σω θα πρέπει να έχουμε ένα μόνιμο εισηγητή για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να το διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξή μα. Και υπάρχει και ένα θέμα ακόμα που ανέφερε η κυρία ε, Τσίμερ. Είναι κάτι το οποίο. Ε, ξέρω ότι έχει συζητηθεί στο ΕΛΚ και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και πάλι για την πολύ καλή δουλειά της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δέβα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τσίμερ για την εξαιρετική έκθεσή της. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λέει, αλλά όσον αφορά την απόδοση της γης ε, είμαι ε, ε, πιο επιθετικός. Καταρχήν διότι πρέπει να υπάρχει νερό και δεύτερον, ακόμη και αν η Σαουδική Αραβία έχει μία μεγάλη έκταση, δεν, δεν μπορεί η επένδυση αυτή να απομακρυνθεί από τον γεωγραφικό της εντοπισμό. Άρα μακροπρόθεσμα ούτως ή άλλως θα εξαρτάται η τύχη αυτής της γης από τις τοπικές αρχές. Και αν οι σχέσεις ε, ε, χαλάσουν τότε το κράτος μπορεί να εθνικοποιήσει και αυτό έχει γίνει διεθνώς σε πολλά μέρη όπως άλλωστε στη Σρι Λάνκα όπου κατάσχεσαν και εθνικοποίησαν τη δικιά μου έκταση. Αυτό λοιπόν ανησυχεί πολύ κόσμο. Όντως έχασα 4.000 ε, εκτάρια, Οπότε το κράτος πάντως, πάντοτε μπορεί να εθνικοποιήσει και οι ξένοι δεν μπορούν να απομακρύνουν τη γη τους. Άρα η ευθύνη του ιδιοκτήτη ε, ουσιαστικά εξαρτάται από τις εθνικές αρχές εκτός εάν κάποιος ε, θέλει να στείλει ένα στρατό να βάλει ένα ηλεκτροφόρο σειρματόπλεγμα ε, πράγματα που έχουν γίνει δηλαδή. Αλλά και αυτά τα μέτρα είναι υπερβολικά. Ε, οπότε, ασχέτως του ποσού που έχετε επενδύσει σε μία έκταση μπορεί το κράτος με δύο γραμμές σε δύο αράδες να το εθνικοποιήσει. Δεν θέλω βέβαια να τονίσω αυτή την πτυχή αλλά κατά τα άλλα πιστεύω ότι είναι εξαιρετική έκθεσή σας. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Όλτοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ε, από την πλευρά της Επιτροπής ε, χαιρετίζουμε την έκθεση της κυρίας Τσίμερ, η οποία είναι καλή και χαιρόμαστε διότι πολλά από τα θέματα που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνονται και σκέφτομαι εδώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει προτεραιότητα σε ορισμένους τομείς, ότι πρέπει να περιλάβουμε ε, το δικαίωμα για διατροφική ασφάλεια ε, και όχι μόνο από πλευρά γεωργική. Αλλά δεν έχουμε εξετάσει εδώ τη ρίζα του κακού σχετικά με την, ε, ε, την διατροφική ασφάλεια και θα ήθελα ε, να το γνωρίζω, αλλά αυτό το λέω εκ του περισσού. Θα περιοριστώ σχετικά με την έκθεση σε τέσσερα θέματα. Καταρχήν, στη σχέση της διατροφικής ασφάλειας σε συνδυασμό με την διατροφική κυριαρχία όπου η συγγήτρια χρησιμοποιεί έναν ορισμό. Εμείς πάντοτε μιλάμε για διατροφική ασφάλεια για κάποιο λόγο διότι η διατροφική ασφάλεια είναι ένας όρος ο οποίος αναγνωρίζεται διεθνώς όλοι ξέρουν περί τίνος ομιλούμε πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την διατροφική κυριαρχία δεν υπάρχει ε, μία σαφής ε, άποψη, δεν υπάρχει ένας ε, σαφής ορισμός και γι' αυτό δεν υπάρχει και άμεση διασύνδεση μεταξύ της διατροφής και του δικαιώματος προς διατροφήν. Δεύτερο θέμα από πλευρά ισότητας των φύλων αναφέρεται στην έκθεση ότι δεν έχουμε δώσει επαρκή προσοχή στην ισότητα των φύλων, πράγμα το οποίο ίσως είναι σωστό και η ισότηση είναι πολύ σημαντική για τη διατροφική ασφάλεια όχι μόνο σε σχέση με τη γεωργία όπου στις υποανάπτυξη χώρες έχουμε πάρα πολλές γυναίκες γεωργούς ορισμένες ε, μάλιστα χώρες είναι η πλειοψηφία αλλά ε, και όσον αφορά την ε, κατανομή των περιουσιακών στοιχείων ε, εντός της ε, οικογενείας βλέπουμε ότι η ισότητα των φύλων είναι πολύ σημαντική και από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε το ε, γεγονός αυτό και γι' αυτό ευχαριστώ την εισηγήτρια που μας το τόνισε. Το τρίτο είναι το θέμα της γης και έχω να κάνω μία σύντομη διόρθωση. Στο σημείο 17 της εκθέσεως της εισηγήτριας το θέμα αναφέρεται κάπως διαφορετικά και ε, ε, υπάρχουν οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την διαχείριση της γης και την δασοκομεία και τέλος ε, υπάρχει ε, ένας διαχωρισμός μεταξύ του εθνικού και διεθνούς επίπεδου και βλέπουμε εδώ όλες τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εφαρμόζονται για την Αφρική, ε, ε, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΦΑΟ που πρέπει να, ε, να προσαρμοστούν σαν εθνικά δεσμευτική νομοθεσία και το, οι δεσμευτικοί κανονισμοί είναι κάπως διαφορετικοί. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έναν σαφή τρόπο με τον οποίο να προχωρήσουμε και θα ήθελα αυτό να σας το επισημάνω. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ε, διακυμάνσεως των τιμών που είναι πολύ σημαντικό διότι τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχε μία μία αναμόρφωση ε, της ε, εκθέσεως που ζητήθηκε από τον πρόεδρο των G20 ε, για να διατυπωθεί η πρόταση σχετικά με το τι γενέστε με την υπερβολική αστάθεια των τιμών των τροφίμων. Και εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο εις την κερδοσκοπία διότι Σύμφωνα με την εισηγήτρια νομίζω ότι λέει ότι η αστάθεια των τιμών οφείλεται στην κερδοσκοπία. Πρέπει εδώ να διαφοροποιηθούμε διότι όντως υπάρχουν ε, διάφορες λειτουργίες ε, όπως οι προθεσμιακές αγορές ε, για να μπορέσει κανείς να λειτουργεί στην αγορά σωστά αλλά η η συμμετοχή ορισμένων εμπλεκομένων διαφέρει από τους εμπόρους των πρώτων υλών και εδώ πρέπει να δημιουργηθεί το σωστό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όντως καταρτίζουμε τέτοιες προτάσεις με πληροφορίες για την διαφάνεια, για την ρύθμιση των αγορών χωρίς όμως να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την διακύμανση των τιμών και ε, πολλά θέματα ε, άπτονται των, ε, της κατάστασης της αγοράς και η κερδοσκοπία υπάρχει όταν μια αγορά είναι στενή και όταν υπάρχει μεγάλη δεν μπορεί κανείς να προβλέψει σωστά ποια εξέλιξη θα υπάρξει και αυτό αντικατοπτρίζει την τωρινή διακύμαση των τιμών που έχει σχέση και με τους περιορισμούς των εξαγωγών. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ε, και να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιους συναδέλφους και εταίρους ανά τον κόσμο μπορούμε να συνεργαστούμε και να αποφύγουμε ε, να κλείνουν τα σύνολα. Τέλος, όσον αφορά τα σιτηρά και τα αποθέματα στον τομέα αυτό που παρουσιάζουν διακυμάνσεις τιμών, ε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αποθέματα αυτά επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά και στο παρελθόν ε, είδαμε ότι ήταν ε, αποτελεσματικά τα μάτρα που ελήφθησαν. Υπήρχε πολιτική παρέμβαση ε, και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αυτά ήταν μερικά από τα θέματα, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, χαιρετίζει η Επιτροπή την έκθεση αυτή και πιστεύουμε ότι έχει πολλά θετικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσίμερ για να ολοκληρώσετε τη τελική φάση. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, πολλές υποδείξεις τις οποίες μου κάνατε και ελπίζω ότι στην Επιτροπή θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το θέμα. Το είπα άλλωστε και στην αρχή κύριε Ντέβα, δηλαδή ότι σε ορισμένες απαιτήσει σαν το land grabbing που ε, ε, ε, έχω ίδιες απόψεις προσπάθησα να είμαι μετριοπαθής για να υπάρξει ευρεία συνένεση. Άλλα θέματα θα προσθεθούν στη συνέχεια. Προσβλέπω και ε, στην ε, ακρόαση η οποία θα γίνει. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και παραδείγματο χάρη θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συζητήσουμε αν σε σχέση με την διατροφική ασφάλεια και το δικαίωμα για διατροφή και τροφή μπορούμε να παραμείνουμε και την γεωργική ε, πολιτική και να δούμε ε, αν ε, επαρκεί οι απαγορεύσεις που υπάρχουν και δεν πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γίνει ανά τον κόσμο αν γεωργοί παράγουν πρώτε ύλες και τελικά αμείβονται ανεπαρκώς για το κόστος της παραγωγής τους. Δηλαδή σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει μία χρηματοδότηση η οποία υπολείπεται του κόστους παραγωγής. Αυτό το οποίο ναι, γίνεται και η διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Διεθνούς Αγοράς είναι ότι έχουμε τις αντισταθμιστικές εισφορές εις ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στις επιδοτήσεις των εξαγωγών για τις υποανάπτυξη χώρες οπότε ε, πρέπει να, ε, να συνεπιφέρουμε και τη συζήτηση της αναμορφώσεως της κοινή γεωργική Πολιτική, διότι όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές γεωργική, ενεργειακή και άλλες οι οποίες εμπλέκονται θα πρέπει να τις συζητήσουμε και γι' αυτό χαίρομαι ότι συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπολογίζει ότι σε θέματα όπως η στήριξη των γυναικών σε όλους τους τομείς το γυναικών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην γεωργία θα ήταν καλή και θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική που θα μπορούσε να επεκταθεί και να καλύψει αυτές ε, τις ε, παραλήψεις με τρόπο ικανοποιητικό. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση της ε, ΦΑΟ, πρέπει να πω ότι στην αρχή της εκθέσεως αυτό στην αρχή αναφέρεται ε, σωστά δηλαδή μπορεί μέσα στο κείμενο να το έχω αναφέρει περιληπτικά αλλά στην εισαγωγή αναφέρω τον πλήρη τίτλο και όσον αναφορά την αστάθεια πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την αστάθεια των τιμών αλλά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να μειώσει την αστάθεια στον τομέα των τιμών και γι' αυτό πιστεύω ότι η δικιά μου θέση διαφέρει από αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να δούμε πώς θα την αξιολογήσει η Επιτροπή μας. Θα παρακαλούσα ε, να συνεργαστούμε για τη διατύπωση των τροπολογιών. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ε, είναι 20 Ιουνίου, 6 το απόγευμα και 13 Ιουλίου θα γίνει η ψηφοφορία. Ε, φτάνουμε τώρα στην πραγματική στρατηγική για τις πρώτες ύλε. Πρόκειται για μία έκθεση της ΙΤΕ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που είναι παραγωγή πρώτων Ο εισηγητής της ΙΤΡΕ είναι ο κύριος Μπουτιγόφερ και θα ήθελα να δώσω το ε, λόγο στην κυρία Σνίπερ Γιάστραμ ε, που είναι η συντράκτη Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Όπως ακριβώς το είπατε, μέχρι το 2050 θα υπάρχει μία αύξηση ε, κατά 314% για την ζήτηση ε, πρώτων υλών. Η έκθεση του κυρίου Βιτιχόφερ νομίζω ότι είναι σωστή ε, και εμείς θεωρούμε ότι διάφορα θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη περισσότερο. Καταρχήν η πολιτική συνεκτικότης, κατά δεύτερον λόγον μία εναλλακτική η λύση στο ισχύο σύστημα των ε, δασμολογικών προτιμήσεων, ένας έλεγχος ε, των μηχανισμών, ε, η αίτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει μία μελέτη της διαφανείας είναι ένα τεράστιο θέμα επί του οποίου θα μπορούσε κανείς να πει πολλά περισσότερα και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ορισμένα θέματα παρελήφθησαν αλλά θα μπορούσαν ε, στις τροπολογίες να συμπεριληφθούν όπως παραδείγματος χάρη το γεγονός ότι ε, μέτρα που αναφέρονται εις ε, την ε, πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε είναι πολύ δύσκολη και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχουν σωστές συμβάσεις δηλαδή δίκες μακροπρόθεσμα εφικτές συμβάσεις για τις πρώτες ύλε, διότι υπάρχουν συγκρίσιμες ε, ε, ε, παρομοιώσεις με το εμπόριο των διαμαντών στην Βοτσουάνα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν διαβουλεύσεις και να προσπαθήσουμε να πείσουμε την αφρικανική πλευρά να ενισχύσει την σκοπιά των πρώτων υλών. Ε, άλλωστε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κίνα στον τομέα αυτό ε, δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία αυτή και υπάρχουν δηλαδή πολύ μεγάλες χώρες οι οποίες μπορεί να έχουν αποκλειστεί. Όσον αφορά την συμφωνία θα πρέπει ε, εδώ ε, να ε, κοιτάξουμε πόσο θα διαμορφωθούν οι ε, δαπάνες ε, και αν στηρίζει κανείς με μία ενίσχυση ε, μία πρώτη ύλη θα πρέπει να έχουμε αξιολογήσει πόσο σημαντική είναι για τη χώρα για την ανάπτυξή της ή για ένα ίδρυμα διότι οι δαπάνες αυτές οι οποίες αναφέρονται στην προώθηση ε, είναι εύκολο να υπολογιστούν. Πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για αξιοποίηση εντός της χώρας και έχουμε τέτοιες συμφωνίες για την επεξεργασία ε, μεταξύ του Καζακστάν και της Γερμανίας ή ε, άλλων περιπτώσεων για να υπάρχει πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Ουσιαστικά όμως βλέπουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια προς όφελος της οικονομίας και να ε, χρησιμοποιήσουμε πρωτοβουλίες σαν ε, την χάρτα των πρώτων υλών ε, και να λάβουμε υπόψη μας και την επανεθνικοποίηση ή την αξιοποίηση σε επικοδομητική συνεργασία. Σερβία. Επιπλέον πρέπει να θεωρηθεί ότι ε, το έργο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί μακροπρόθεσμα και σε πολύ γενικές γραμμές διότι εδώ δεν θέλαμε να θίξουμε καμία βιομηχανία αλλά είναι δύσκολο ε, ε, να, να γίνει αυτό για 12 στρατηγικές πρώτες ύλες. Προσλέπω εις τις τροπολογίες που η προθεσμία θα λήξει σε δύο μέρες, δηλαδή στις 26 Μαΐου. Κύριε Κυρία Σαρζεντίνη, έχει λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την ε, γνώμη αυτή. Στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ασχοληθήκαμε με τις πρώτες ύλες και είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι αρκετές επιτροπές ασχολούνται με το σημείο αυτό και αυτό είναι κάτι το θετικό. Έχει να κάνει με όλες τις βιομηχανίες της Ευρώπης και τις γεωπολιτικές σχέσεις στον κόσμο. Έχει να κάνει και με τις αναπτυσσόμενες χώρες τόνισε η συγγήτρια ορισμένα σημεία και η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε μερικά από αυτά τα σημεία με τη σειρά μας να ενισχύσουμε και μετά να φτάσει αυτή η γνωμοδότηση στην Ήτρε και να μπορέσει να βελτιώσει την ιδεγία για τις πρώτες ύλες στην Επιτροπή αυτή. Έτσι βελτιώνεται η όλη συζήτηση μπορούμε να πούμε εκείνο που επιθυμούμε εμείς και να μιλήσουμε για τη διαφάνεια, το ένα το άλλο, αλλά πρέπει σε τελική ανάλυση να φτάσουμε σε μια πρόταση για να μπορούμε να παρουσιάσουμε και να συνδυάσουμε με εκείνη των υπολείπων επιτροπών. Εδώ δεν πρόκειται να αλλάξουμε μερικά πράγματα εδώ και εκεί, να αντιγράψουμε αυτό που ήδη η Κίνα κάνει σε αυτό. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση, κάτι το πιο τίμιο, μια πολιτική ας πούμε επενδύσεων και θέσπισε το Κοινοβούλιο τώρα πρόσφατα, μάλλον συνέταξε ένα κείμενο, το υιοθέτησε για την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες σε αρκετές χώρες ε, για τους επενδυτές. Χρειάζεται λοιπόν μία συνοχή στην πολιτική αυτή. Στο άρθρο 1 Εντάξει, καλό. Ίσως όμως θα μπορούσαμε να είμαστε και περισσότερο σαφείς σε αυτό το άρθρο 1. Και ακόμη κάτι. Όχι για τις εξαγωγές. Να πούμε ότι μία χώρα που δεν ε, παίρνει φόρους, ε, τότε θα πρέπει να επιβάλλει φόρους και δασμούς σε άλλα προϊόντα, στο ενόπνευμα, στον καπνό κλπ. Λοιπόν, για τις πρώτες ύλες να υπάρχει υψηλότερες ε, φόρους ε, για παράστα ή μη κατεργασμένα προϊόντα, γιατί αυτά μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίες και χρειάζεται ένα κείμενο για τις πρώτες σύλλε ώστε μια χώρα να μπορεί να αναπτυχθεί κατάλληλα. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε χώρες ε, που είναι σε ένοπλη σύραξη λόγω του πλούτου τους να συνεχίσουν να ρυθμίζουν πράγματα με τον τρόπο αυτό. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είναι εδώ και οι συνάδελφοι που εκπροσωπούν ε, την Γενική ε, Διεύθυνση Βιομηχανίας. Θα ήθελα να κάνω μερικές συστάσεις για τις προτάσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Δεν έχω ιδιαίτερες αντιρρήσεις, όμως κάποιες διευκρινήσεις ενδεχομένως. Για το πρώτο θέμα, Μιλάω για την ε, συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Συμφωνώ απόλυτα και θα έλεγα ότι η ανακοίνωση η οποία σας υπευλήθη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ήδη μια συγκεκριμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σαφές ότι μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης Λισαβόνας ε, η συνοχή της ε, αναπτυξιακής πολιτικής είναι όχι μόνο μια καλή αρχή πολιτικής, αλλά είναι και μια υποχρέωση νομικής ε, φύσεως. Όσον αφορά το GSP, το Γενικευμένο Σύστημα Προεδημήσεων, μπορώ να σας καθησυχάσω. Λίγες πρώτες ύλες ε, εκτός του γεωργικού τομέα υπόκεινται σε ε, τελωνιακούς δασμούς ε, και μιλάω κυρίως για πρώτες ύλες μεταλλευμάτων και, μεταλλευμάτων και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και δύο-τρεις εβδομάδες ενέκρινε ένα, για το, ένα ε, πρόγραμμα για το GSP μετά το 2014 που δεν ε, ε, προβλέπει ιδιαίτερες αλλαγέ για τα προϊόντα που καλύπτονται. Υπάρχουν κάποιες καινοτομίε, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με την κάλυψη των προϊόντων που ήδη καλύπτονται από το σύστημα αυτό. Αυτό σας το λέω ε, στο πλαίσιο της ανακοίνωση που υποβάλαμε προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα τη διαφάνεια, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. και στην ανακοίνωσή μας, όπως και στην προηγούμενη του 2008, είναι σαφής η υποστήριξη για την διαφάνεια της, ε, ε, του κλάδου των μεταλλευμάτων γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές από την νομοθεσία Dot Front ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς θέλουμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία αυτή στο πλαίσιο προτάσεων που έχουν δρομολογηθεί για τη διαφάνεια ε, των ε, συναλλαγών των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών και όσον αφορά το reporting ε, αναχώρα, αναφέρεται και αυτό στις προτάσεις. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία υπάρχουν κάποιες από τη χρηματοδότηση για την, από την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα και γι' αυτό η ιδέα είναι να υπάρξει μια πολύ στενή και αυστηρή παρακολούθηση που θα είναι κατάλληλη για τα διάφορα προγράμματα. Αυτή τη στιγμή αυτά εγκρίνονται από την ΕΤΕ. Υπάρχει επίσης μια αναφορά στην ε, περιεκτική ανάπτυξη, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, inclusive growth στα αγγλικά. Ο σημαντικότερος ρόλος δηλαδή του νομοθέτη, στην κάτι που θα αναφέρεται στην πράσινη βίβλο για το θέμα ε, αυτό, νομίζω ότι και αυτό πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και όσον αφορά τώρα τις ε, μικρές εκμεταλλεύσεις, τις των ε, ε, μικρότερων μεταλλορυχείων ε, θα έλεγα ότι μία από τις ανησυχίες είναι η διευκόλυνση της μετάβασης από τον άτυπο στον επίσημο τομέα όσον αφορά τις δραστηριότητες των ορυχείων με τις δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα την, ε, τον κατακαιρματισμό, την αποδυνάμωση του συγκεκριμένου τομέα. Και θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, της ε, Συμφωνίας Ισότιμων Συναλλαγών μεταξύ των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, είναι ένας τομέας στον οποίο παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στον οποίο όμως υπάρχουν και άλλοι εταίροι που συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό, όπως για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα που έχει και ένα καταπίστευμα πίστευμα για την ενίσχυση των προσπαθειών στον τομέα αυτό, όπως επίσης η Αφρικανική ε, Τράπεζα Ανάπτυξης και όπως ε, επίσης ε, και η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης μας ζήτησε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό και να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες ενίσχυσης των όσων ήδη υπάρχουν, των ήδη υφισταμένων μέσων. Κάτι ακόμη για, τις, ε, για τους εξαγωγικούς φόρους. Γνωρίζετε ότι δεν την χάνουν ιδιαίτερη υποστήριξη σε πολλούς τομείς, ε, δεν είναι πολύ δημοφιλής και δεν είναι πάντοτε και συμβατές με τις υποχρεώσεις ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις, αλλά όλοι οι οικονομολόγοι της ανάπτυξης συμφωνούν ότι υπάρχουν πιο αποτελεσματικά μέσα τα οποία μπορούν ε, να επιφέρουν καλύτερη διαφάνεια και δημοσιονομικά αποτελέσματα καλύτερα για τις ε, αναπτυσσόμενε χώρε. Βέβαια αυτό σημαίνει μεταρρυθμίσεις που δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνουν σε χώρε οι οποίε έχουν κάποια όρια σε ζητήματα διακυβέρνηση. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να ζητήσω από το συνάδελφο τη Γενική Διεύθυνσης Βιομηχανία, αν μου δίνετε το λόγο, να αποσαφηνήσει κάποια από τα ζητήματα που ενδεχομένω να ξέχασα. Δεν... Όχι, δεν είχε προβλεφθεί γι' αυτό σύντομα, σύντομα, σύντομα από τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων. Ε, εγώ είμαι ο συντονιστή για τις ε, πρώτες ύλες για το θέμα αυτό, για την ανακοίνωση αυτή. Ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος, θα ήθελα κάτι απλώς να τονίσω εκτός από τις γενικέ αρχές και είχε τη δυνατότητα ήδη να εξηγήσει κάποιες από τις αρχές αυτές, ε, εγώ παρακολούθησα κάποια από τα σχόλια ε, των προλαλισσάντων, των ε, ευρωβουλευτών, πρέπει να περάσουμε από τις γενικέ αρχές σε συγκεκριμένε δράσεις. Γι' αυτό ακριβώ. αυτό μα ζητούν στι επαφέ μα οι αφρικανικές χώρε. Δηλαδή, το το αφρικανικό όραμα για τα ορυχεία, για παράδειγμα. Θέλουν ένα συγκεκριμένο χάρτη πορεία και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να του υποστηρίξει σε κάποιε από αυτέ τι δράσει του. Έχουμε τώρα μια συγκεκριμένη συμφωνία. Έχουμε μια συγκεκριμένη συμφωνία ε, την οποία, ε, την οποία ε, υπογράψαμε ε, με την Αφρικανική Ένωση, ειδικότερα για ε, τα ορυχεία και καλύπτει την καλή διακυβέρνηση, τις δεξιότητες και τις ε, γεωλογικές γνώσεις. Έχουμε λοιπόν το πλαίσιο, έχουμε την πολιτική θέληση και υπάρχει και μία ευθύνη από τη δική μας, στη δική μας πλευρά. Πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε και ζητώ από το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει. Έχει να κάνει και με κάποια από τις παρεμβάσεις κάποιου ευρωβουλευτή. Ε, η οργάνωση δηλαδή ενός εργαστηρίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Αφρικανικής Ένωσης ε, για τα τελειωνία. Οπότε πάρα πολύ θα μας ευχαριστούσε αν υπήρχε στην έκθεση μία αναφορά για την συνεργασία αυτή, για τη Συμφωνία Συνεργασίας για τις πρώτες ύλες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής ε, Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κυρία, θέλετε να παρουσιάσετε τα συμπεράγματα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι τοποθετήθηκαν. Όπως σας είπα έχουμε προθεσμοί για τις τροπολογίες μέχρι τις 26 Μαΐου και πιστεύω ότι δεν θα ήταν κακό να υπάρξουν ορισμένες συμπληρώσεις. Ε, ε, τώρα όποιος ε, και να έχει διατυπώσει γνωμοδότηση είτε η Ήτρε είτε άλλες επιτροπές ε, πιστεύω ότι όλοι συμπλέουμε προς τον ίδιο στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία είναι μέχρι 26 Μαΐου το μεσημέρι και θα ψηφίσουμε 14 Ιουνίου. Αυτό οφείλεται στο λόγο ότι πρέπει να έχουμε ψηφίσει πριν από τις 30 Ιουνίου και πριν καλυφθεί η ημερομηνία για τις τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν ε, τώρα ε, ένα άλλο θέμα. Έχουμε ε, την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες όπου υπήρξε μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντέβα ο οποίος προείδρευσε για να παρουσιάσει τα πορίσματά του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Διακόπτη η Πρόεδρος, παρακαλώ λίγο ήσυχα να αποχωρείτε. Κυρία Πρόεδρε, αυτή η αποστολή στη, στον ΟΗΕ, αυτή η τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Θεοχάρους, την Κορίν Κρέτσου, ε, που με βοήθησαν. Είχαμε μια πάρα πολύ έντονη, ε, ένα πολύ ε, φορτωμένο πρόγραμμα. Είχαμε μάλιστα και ιδιαίτερη βοήθεια από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω. Βέβαια δεν είναι όλοι εδώ. Είχαμε μία σειρά συναντήσεων, αλλά πριν ε, πάμε στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, ε, ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο ότι δεν θα δεχθούμε να μας μεταχειριστούν ως συμβούλους και ότι θέλουμε να παίξουμε έναν πλήρη ισότιμο ρόλο στις ε, εργασίες του ΟΗΕ. Θέλουμε να είμαστε ισότιμοι με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ζητήματα αυτά και μας δόθηκε κάθε εγγύηση από τον ε, Επίτροπο ότι έτσι όντως θα μας συμπεροφέρονταν. Και όντως αυτό συνέβη. Θα ήθελα μάλιστα να αναφερθώ στο εξής και θα ήθελα επισήμως να αναφερθεί το τι συνέβη με τον κύριο Πίμπαλξ έκανε τεράστιες προσπάθειες για να, μπορέσει, για να μπορέσουμε να είμαστε ισότιμοι στην όλη διαδικασία με τους υπόλοιπους και να μην είμαστε ε, ε, δεύτερης κατηγορίας για να το πω έτσι. Είχαμε πρόσβαση στην Ολομέλεια, είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε όποιον θέλαμε, ε, πήγαμε σε όλα τα εργαστήρια και ήμασταν ε, πλήρη, συμμετείχαμε πλήρως ε, σε όλες τις ε, δραστηριότητες. Οπότε θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί κατάλαβε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια δημοκρατική διάσταση, ένα δημοκρατικό στοιχείο, ειδικότερα όταν μιλάμε για τα λεφτά των φορολογουμένων. Τώρα, γιατί οι χώρες αυτές είναι σημαντικές. Πριν από 10 χρόνια σε αυτήν την Επιτροπή εγκρίναμε το anything but arms, οτιδήποτε εκτός από όπλα που σκοπό είχαν να βοηθήσει τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να περάσουν οι χώρες αυτές από λιγότερο ανεπτυγμένες σε κάπως πιο ανεπτυγμένες. Όμως μετά από 10 χρόνια μόνο δύο χώρες έχουν κάνει τη μετάβαση αυτή και οι υπόλοιπε έχουν ε, παραμείνει στην κατάσταση που ήταν. 48 χώρες ε, είναι, ο αριθμός είναι σήμερα απαριθμώνται μεταξύ των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και ε, δημιουργούμε ένα μηχανισμό για να, τους, ε, να τις διευκολύνουμε να ε, κάνουν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, χωρίς περιορισμούς και το, το αποκαλούμε αυτό anything but arms, οτιδήποτε εκτός από όπλα. Βέβαια, έχουμε κάποιους περιορισμούς στο τι μπορούν να εξάγουν και να γίνει λοιπόν το anything but arms, anything but farms. Δηλαδή ε, οτιδήποτε εκτός από όπλα να γίνει ε, ε, οτιδήποτε εκτός από αγροκτήματα, γιατί πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα ε, εξάγονταν. Ελπίζουμε λοιπόν και το γενικό συμπέρασμα είναι ότι θα έπρεπε επόμενες, στα επόμενα 10 χρόνια να φτάσουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες από 48 στις 24 στο ίμιση δηλαδή. Δηλαδή να βελτιώσουμε το ποσοστό μετάβασης των χωρών από τη μία κατηγορία στην άλλη. Πέντε μήνες με διαπραγματεύσεων είχαν ως αποτέλεσμα όχι 0,5 αλλά 0,2 των, του εισοδήματός μας, να, ε, των εσόδων μας, συγγνώμη, να ε, πηγαίνουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Τι να σας πω, κατά πόσο αυτό είναι ιδιαίτερη επιτυχία εξαρτάται από το τι θα κάνουν οι ίδιες οι χώρες αυτές ε, για να βοηθήσουν ε, τους, ε, τους εαυτούς τους να περάσουν από την κατηγορία των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών σε πιο ανεπτυγμένες χώρες. Όμως, ένας κούκο δεν φέρνει την άνοιξη, άρα πρέπει και αυτές οι χώρες να προσπαθήσουν. Εμείς προσπαθήσαμε να ε, τους ζητήσουμε να κάνουν περισσότερες επενδύσεις ε, ε, στην ε, απασχόληση στην ανάπτυξη των φυσικών πόρων, ε, την ανάπτυξη των τοπικών εξαγωγικών τους ε, δυνατοτήτων, ε, ειδικότερα στην γεωργία, στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες. Γνωρίζετε ότι η δυνατότητα μεταποίησης είναι πάρα πολύ χαμηλή, το γνωρίζετε και εσείς κυρία Πρόεδρε, όμως μπορεί να περάσουν από τη γεωργία στις υπηρεσίες. Πολύ πιο γρήγορα από όσο φανταζόμαστε και το έχουμε δει σε ορισμένες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής τη χρήση της κινητής τηλεφωνίας για παράδειγμα, όχι μόνο για υπηρεσίες πληροφόρησης, αλλά και για οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με οικονομικές συναλλαγές, ε, είτε ρευστού, ε, είτε ε, εξέβρεση καλύτερης τιμής για ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι για παράδειγμα η πρόσβαση στις ήταν κάτι το πάρα πολύ θετικό γιατί δίνει τη δυνατότητα στις χώρες αυτές ε, να κάνουν τη μετάβαση στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης ενθαρρύναμε τις χώρες αυτές και ο Επίτροπος Μπίλβαρς είναι αποφασισμένος να το κάνει αυτό, να ισχύσει ακόμη περισσότερο τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, στην μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειων. Επίση, ζητήσαμε από τι χώρε αυτέ να άρουν οποιαδήποτε εμπόρια υπάρχουν για τι επενδύσει, ώστε ξένοι επενδυτέ, να μπορούν να είναι ομοχλός τη ανάπτυξη, κάτι που θα βοηθήσει στη μετάφαση των χωρών αυτών σε πιο ανεπτυγμένες χώρες, από τη στιγμή βέβαια που έχουν την κατάλληλη νομική βάση, από τη στιγμή που υπάρχει ασφάλεια για τις υποδομές, υπάρχει επιβολή των συμβολέων που συντάπτουν, συνάπτονται πνευματικά δικαιώματα και νομικώς δεσμευτικές ε, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτά είναι ε, ανάπτυξη θεσμών ουσιαστικά, αποτελούν ε, ε, ανάπτυξη θεσμών, όμως πρέπει για να τις βοηθήσουμε να δεχθούν τις δικές μας απαιτήσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών μας. Εν δηλαδή, ήταν πάρα πολύ πάρα πολλέ ε, και επικοδομητικές οι συνεδριάσει στις οποίες συμμετείχαμε και είχαμε την εντύπωση, τουλάχιστον έτσι αναφερόταν γραπτός, ε, σε πολύ επικοδομητικές ε, προτάσεις όσον αφορά τη σχέση μας, τη συνεργασία μας με τις χώρες αυτές στα επόμενα χρόνια. Το θέμα όμως εξαρτάται από το πώς θα ενεργήσουμε και σε τι χρονικό ορίζοντα. Επίσης, ε, περίπου 50 αρχηγοί ε, κρατών στην Ολομέλεια, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Ιράν, που από ό,τι κατάλαβα δεν είχε καταλάβει τίποτα, ούτε είχε ακούσει τον Άνταμ Σμιθ ποτέ, γιατί συνέκρινε χώρες ε, οι οποίες βγάζουν ε, λεφτά, παίρνοντας λεφτά από φτωχές χώρες και δεν, έχουν ε, την, δεν έχει την παραμικρή σχέση νομίζω με την οικονομία και με την, ούτε καν με την γένεση του κόσμου για να το πω έτσι και ίσως θα έπρεπε να του στείλω ένα γράμμα να του εξηγήσω πώς ακριβώς έγινε αυτό Εν πάση περιπτώσει, Οι τουρκικές αρχές ε, ήταν πραγματικά πολύ φιλόξενες, ε, ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τα θέματα ασφαλείας και ήταν πάρα πολύ ε, ανοιχτές στα αιτήματά μας για πρόσβαση ε, σε όλες τις συνεδριάσεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ε, πω και πάλι ότι είμαι πολύ ευγνώμων και στους συναδέλφους για όλη τη δουλειά που έκαναν εκ μέρους Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα. Κύριε Κρέτο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους μου και τις συναδέλφους από τη Γραμματεία που μας στήριξαν και όντως ήταν μια εξαιρετική συνεδρίαση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρόλο που τέθηκε το θέμα της αποτελεσματικότητας αυτών των συνεδρίων που οργανώνονται κάθε 10 χρόνια και συγκεντρώνουν άτομα με πολύ υψηλούς στόχους και μετά βλέπουμε ε, μετά από τρεις δεκαετίες τέτοιων ασκήσεων ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιζητουμένων στόχων και της ε, πραγματικότητας ε, και πιστεύω ότι αυτές οι συνεδριάσεις θα πρέπει να οργανώνονται στα πλαίσια του ΟΗΕ για να είναι πιο αποτελεσματικές. Υπήρξαν πολλές δραστηριότητες, αλλά για μένα είναι σαφές ότι ε, πρέπει να αναγνωρίσει κανείς τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που συμβάλλει στην διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στις συζητήσεις μας με ε, τον ε, Επίτροπο Πίμπαλς, ο οποίος ε, ήταν διαθέσιμος και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε για την προθυμία του και τη συνεργασία, αλλά πρέπει ε, να ξέρουμε ότι ε, υπήρξαν και ακραίες θέσεις, όχι μόνο ο κύριος Τζάντα, αλλά πολλοί επέπληξαν τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες για την κατάσταση τους και Ε, ε, υπήρξε μία δυσαρέσκεια αλλά βέβαια φοβάμαι ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και πιο σοβαρές κρίσεις Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, για το πώς διαχειριζόμαστε αυτή την πολιτική διάσταση και θα πρέπει να γίνει και άλλη μία συζήτηση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Και στην ε, πόλη είχαμε μία τέτοια ε, συνεδρίαση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προωθήσουμε τέτοιες ε, πρωτοβουλίες από επιτροπές και αναλλαγές. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά από όσα έχουν πει και ο κύριος Δέβα και η Κορίνα, εγώ ελάχιστα έχω να προσθέσω. Οι συζητήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους των υποαναπτύκτων των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, των φτωχών χωρών, αλλά και με τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μας έχουν πείσει ότι πραγματικά χρειάζεται εξαγωγή, επιτρέψτε μου τον όρο, δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτές τις χώρες. Δηλαδή είναι πρότιστο καθήκον να εμπεδώσουμε, να εδραιώσουμε την δημοκρατία, την σωστή διακυβέρνηση, τα δημοκρατικά Ινστιτούτα σε αυτές τις χώρες και να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση γιατί υπάρχει διαφθορά σε πολλά επίπεδα και μόνο αν παρακάμψουμε αυτή τη διαφθορά και μπούμε κατευθείαν στην κοινότητα και αυτό μας το λένε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα μπορέσουμε να έχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας μηχανισμός παρακολούθησης της εξέλιξης, δηλαδή να μην το αφήσουμε για μια πενταετία ή μια δεκαετία χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Άρα πρέπει, ε, ε, έχει, εκπονηθεί ένα πρόγραμμα. Την εφαρμογή αυτού του προγράμματος πρέπει να την ε, ναι, παρακολουθούμε και να ξέρουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα τελειώσω λέγοντας ότι πολύ σωστά ήταν παρόν εκείνο ο εκπρόσωπος του Ιράν, ο πρόεδρος του Ιράν και τόσες δεκάδες άλλοι αρχηγοί κρατών, υπουργοί εξωτερικών. Επισημαίνω όμως και το είχα επισημάνει και πριν τρεις μήνες ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν εκεί, δεν προσεγκλήθησε καμία εκδήλωση γιατί η Κύπρος δεν είχε προσκληθεί σε αυτή την εκδήλωση. Από την χώρα που διοργάνωνε το γεγονός αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να κάθεται έξω από το επίσημο γεύμα, από το επίσημο δείπνο ο Υπουργό Εξωτερικών μίας από τις 27 χώρες. Δεν ξέρω σε τι ενέργειες προέβη η Επιτροπή, ωστόσο νομίζω ότι για να είμαστε σε θέση να εξαγάγουμε δημοκρατία πρέπει να σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τη δημοκρατία και αν μια χώρα θέλει να λέγεται δημοκρατική και να χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει πρωτίστως να σέβεται τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Κύριος Βίλκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ε, θερμές φιλοφρονήσεις για τον ε, Επίτροπο Πίλμπαξ και θα του τα μεταβιβάσω. Πρέπει εδώ να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα από την παρουσίαση του κυρίου ο ε, το συνέδριο και ένα από αυτά ήταν ε, ε, η συνεργασία που ήταν ένα από τα πιο δύσκολα θέματα προς διαπραγμάτευση και το θέμα είναι ότι ε, αμφισβητήθηκε ποιος έπρεπε να βοηθά τις, τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο. Θα έπρεπε να είναι οι κλασικοί δωρητές ή έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι ε, παίκτες εις την διεθνή σκηνή που θα είχαν κάποιο ρόλο να παίξουν. Και αυτό ήταν πολύ ουσιαστικό γιατί τις διαπραγματεύσεις και αν δεν επηρέασε αρνητικά, εν πάση περιπτώσει ε, ήταν προφανής στις συζητήσεις και εις ε, την Κωνσταντινούπολη διαπιστώθηκε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, δεν επρόκειτο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να προχωρήσουν σε τέτοιες συνεργασίες και ε, τώρα υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου κατά τρότον ώστε να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και ε, να μπορέσουν να προχωρήσουν στα επόμενα λοιπόν συνέδρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διατυπώσει τα είδη των συνεργασιών όπου βλέπει ε, να αναπτύξει με τις χώρες αυτές και τέλος ε, το θέμα είναι το πότε θα φτάσουν στο σημείο αυτό και ποια κλιμακωτή διαδικασία πρέπει να υιοθετηθεί. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ε, κοιτούν όλους τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης της Κωνσταντινούπολης και προσπαθούν να την ε, εφαρμόσουν όσο καλύτερα μπορούν σε συνεργασία με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει μία τάση των μη ανεπτυγμένων χωρών οι οποίες δεν θέλουν να προωθηθούν διότι θα χάσουν ορισμένα από τα προνόμια εγκαταλείποντας τη θέση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Γι' αυτό και εις ε, το συμπέρασμα της Κωνσταντινούπολης υπάρχει ε, μία πρόταση ε, για το Συμβούλιο του ΟΗΕ να υπάρξει μία ομαλή βαθμία αναβάθμιση η οποία θα θεωρηθεί σαν βέλτιστη πρακτική για όλους τους τομείς εκτός από τους οπλισμούς κατά ώστε οι χώρες αυτές να μπορέσουν να βοηθηθούν και να προχωρήσουν στον τομέα αυτό. Αλλά θα πρέπει επίσης πέραν αυτού να εξετάσουμε και άλλα θέματα τα οποία θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές να αναβαθμιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι γενικώ η προσπάθεια αυτή δεν ήταν και αμυγός επιτυχής. Έγιναν πολλές συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα κατάφερε ε, γιατί υπήρχε υψηλή συμμετοχή από τον κύριο Μπαρόζο με τους επιτρόπους Πίμπαλς και Ντεχούχτ ε, αλλά το τελικό έγγραφο θα μας δείξει πόσο στο μέλλον θα μπορέσουμε να ε, έχουμε πιο ισοσκελισμένα έγγραφα τα οποία θα μπορέσουν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να υιοθετηθούν ομόφωνα. Κάτι που δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία σε αυτές τα συνέδρια και αυτό άλλωστε ήταν κάτι που είπαν και διάφορα άλλα κράτη-μέλη. Κύριε Ντεβά, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ναι, γνωρίζω ότι περνάει και ο χρόνος. Ένα θέμα η σε συνάδελφο, το οποίο πιστεύω ότι θα ήθελα να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα κοιμόμαστε τα επόμενα δέκα χρόνια όταν θα αναθεωρούμε την κατάσταση και θα βλέπουμε πώς πάνε οι προσπάθειές μας κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Ευχαριστώ πολύ λέει ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Το, ερώτημα, το πρόβλημα που υπάρχει με την αναπτυξιακή συνεργασία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι ότι δεν είναι μία ομάδα χωρών ε, ε, στις οποίες επικεντρωνόμαστε κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών πολιτικών ή δράσεών μας. Το κάνουμε για το εμπόριο, γιατί υπάρχει ο ΠΟΕ, αλλά επειδή οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες δεν είναι μία ομάδα που αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα ή ε, άλλους οργανισμούς. Ε, ήταν περιορισμένη η προσοχή που, τις, ε, που τους δίναμε μέχρι τώρα σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία εννοώ. Όμως βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές προσπαθούμε να τα πλαισιώσουμε βάσει των διαδικασιών του ΟΗΕ και των ετοιμάτων των απαιτήσεων από πλευρά ΟΗΕ. Κάτι το οποίο ευχαρίστω να μοιραζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτικά. Η διαδικασία παρακολούθησης ε, και συνέχισης αυτού του προγράμματος ε, της ε, Κωνσταντινούπολης είναι κάτι το οποίο πρέπει ακόμη να αποσαφινιστεί περισσότερο στις λεπτομέρειές του αλλά είναι κάτι το οποίο θα δούμε και στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση που θα κάνουμε το 2015. Πριν βέβαια από το 2015 θα πρέπει να δούμε τι έχουμε καταφέρει. Το τι θα κάνουμε λοιπόν πριν από αυτό σε ετήσια ή διετή βάση θα πρέπει να το δούμε, αλλά βεβαίως ευχαρίστως ε, να, σας, ε, να το μεταφέρω το έτοιμά σας. Υπό το DCI, ε, λέει ο κύριος Δέβα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχουμε περισσότερη ε, κάνουμε παρα, ε, μεγαλύτερη ε, αξιολόγηση και παρακολούθηση των στρατηγικών εγγράφων των χωρών αυτών. Μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε περισσότερο, γιατί είναι πραγματικά μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες των χωρών αυτών να είναι τόσο λίγο ανεπτυγμένες. Ε, η Ινδία, η Κίνα, το Βιετνάμ, όταν θα αρχίσουν να είναι σε θέση να μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά θα φτάσει κάποια στιγμή που δεν θα έχουμε πια τίποτε να αναπτύξουμε. Κυρία Θεοχάρους. Από την άλλη, σύμφωνα με δεδομένα που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της διάσκεψης αλλά και προηγουμένως, οι περισσότερες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν εκφράζουν την πρόθεση να περάσουν από τη μία κατηγορία στην άλλη, δηλαδή από λιγότερο ανεπτυγμένες να γίνουν πιο ανεπτυγμένες και αναρωτιέμαι αν χρειάζεται να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος ε, ελέγχοντας κάθε τακτά, κάθε τακτό χρονικό διάστημα, εν πάση περιπτώσει, ε, το τι κάνουν, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμία ελπίδα ανάπτυξη για τις χώρες αυτές. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όχι μόνο να δίνουμε καρότα, αλλά να δίνουμε και μαστίγια. Διαφορετικά, μόνο καρότο θα παίρνουν και γι' αυτό δεν θα περάσουν ποτέ από τη μία κατηγορία στην άλλη. Αν όμως υπάρχει και ένα μαστίγιο, θα το ξανασκεφτούν. Νομίζω ότι είναι ε, θέμα που γρήγορα, γρήγορα θα πρέπει να ασχοληθούμε μαζί του. Γιατί γιατί δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε όλοι όσον αφορά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Θα περάσω όμως στο επόμενο συμπείο. Αυτά. Σήμερα για να ολοκληρώσουμε θα έχουμε την Επιτροπή Παρακολής των Προεδρικών Εκλογών στην ε, Νιγηρία. 16 Απριλίου και πολυάριθμη αντιπροσωπεία υπό την Προεδρία ακριβώ του συναδελφού Πέτερλε, ο οποίος μόλις ήρθε τρεις μήνες, Απρίλιο, και μέχρι και Μάιο και με μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη Μαρία Ντεντέσεβα και τα υπόλοιπα μέλη την του Λαϊκού ήταν ε, με κύρια Λαμπέρ, Λόπεζ Αρκεδάν, Αλγκυλάρ και Μοντάλντο. Να ακούσουμε πρώτα την έκθεση του κύριου Πέτερλε και μετά της κυρίας Νεντέλτσεβα και παρακαλώ όχι πάνω από 3-4 λεπτά ο καθένας τους. Εντάξει, ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερλε πρώτος. Hvala lepa za besedo. Jaz sem vesel, da sem doživel to posebno izkušnjo s sto enainštirideset dolgoročnimi in kratkoročnimi opazovalci. υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα για τη διερμηνία. Ναι, ναι, δεν έχουμε την διερμηνία, έτσι. Ένα, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως μπορείτε να με ενημερώσετε γιατί δεν υπάρχει διερμηνία από τη γλώσσα του μιλητή. Τι δεν υπάρχει ε, διερμηνία, υπάρχει τεχνικό τεχνικό πρόβλημα ή μήπως δεν υπάρχει καθόλου καμπίνα στη γλώσσα μου. Δεν με ενημερώνει κανείς λέει πρόεδρος. δεν αναγνώριζαν τη γλώσσα σας. Ακούτε σλοβενικά τίποτα. Ναι, τεχνικό πρόβλημα λύνεται, είτε ο κ. Πέτερλε θα μας μιλήσει σε, δεν ξέρω σε ποια άλλη γλώσσα. Όχι, δεν υπάρχουν σλοβενικά στην αίθουσα. Υπέροχη μέρα. Ε, συμβαίνει μερικές μέρες έτσι. Μπορείτε να μας τα πείτε στα αγγλικά. Ναι, στα αγγλικά θα συνεχίσω. Και ο συνάδελφος στα γαλλικά. Λοιπόν, ήταν... Ε, ήταν μια πολύ απαιτητική συνάντηση στην Ιγυρία με πολλούς παρατηρητές και ξέρετε ότι ήταν πολύ σημαντική η κατάσταση πριν τέσσερα χρόνια και γι' αυτό είχαν διατυπωθεί και πάρα πολλές συστάσεις και ορισμένες από αυτές ε, όντως ε, ελήφθησαν υπόψη από τις αρχές της Νιγηρίας οπότε ε, άλλαξε το σύνταξαγμα άλλαξε ο ε, εκλογικός νόμος ε, και ε, νομίζω ότι αυτή τη φορά υπήρχε καλύτερη δομή και καλύτερη τοποθέτηση και μπορέσαμε να διασφαλίσουμε ότι τελικά θα υπήρχαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις αν και ξέρετε ότι για τις αρχές Απριλίου ακυρώθηκαν οι εκλογές διότι ε, δεν είχε δοθεί το αναγκαίο υλικό σε όλους τους εκλογικούς ε, σε όλα τα μήματα, τμήματα αλλά διαπιστώσαμε τελικά ότι υπήρχαν 73 ε, εκατομμύρια οι ε, ψηφοφόροι οι οποίοι μπόρεσαν να ψηφίσουν ικανοποιητικά και σε γενικές γραμμές υπήρχε μια καλή ε, ε, εκλογική διαδικασία αργότερα όμως ε, εις τις πιο ευαίσθητες φάσεις υπήρξαν περισσότερα προβλήματα και αυτό περιελήφθηκε στην τελική μας έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί σε μία εβδομάδα στην Αμπούζα. Θα ήθελα να σας πω ότι μετά οι εκλογές πήγαν καλά και μετά από τις τις ε, προεδρικές εκλογές οι ε, κοινοβουλευτικές ε, πήγαν καλύτερα αλλά μετά τις προεδρικές εκλογές υπήρξαν επεισόδια βίας λιγότερα όμως σε σχέση με πρωτετραετίας. Γι' αυτό και πάλι σχετικά ικανοποιηθήκαμε διότι ε, είδαμε ότι υπήρξε πολλή βία ε, αλλά γενικώ η διοργάνωση ήταν καλύτερα από ό,τι προ τετραετίας. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρξε μία Επιτροπή Παρακολούθησης αντελήφθηκα ότι ήταν ικανοποιημένη για την παρουσία μας και είχαμε ένα συντονιστικό ρόλο σε σχέση με τις άλλες αποστολές μπορώ να πω ότι καταφέραμε να διατυπώσουμε και μία κοινή δήλωση και οργανώσαμε συνεδριάσει συντονισμού και το ότι έγινε εκεί αποτελεί μια καλή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Νιγηρίας και πρέπει αυτή η κίνηση να συνεχιστεί. Ε, γι' αυτό και ε, δεν, δεν παράγουμε αυτή την έκθεση για να την παρουσιάσουμε σε δύο-τρεις μήνες, αλλά ήδη τώρα κατά τρόπον ώστε να προχωρήσει η διαδικασία η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή και αντιλαμβανόμαστε ότι ε, όλες οι πηγές έχουν ότι όλες οι εκλογές έχουν ορισμένα ασαφή σημεία ακόμη και πρέπει να υπάρξει και προληπτική δραστηριότητα. Πιστεύω δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να κάνει κάτι συγκεκριμένο στα πλαίσια αυτά. Νομίζω ότι αυτά είχα να σας πω και θέλω να ε, ε, ευχαριστήσω την κυρία Ρέτροβα και τις, τους άλλους συμμετέχοντες σε αυτή την επιτροπή. Νομίζω ότι ήμασταν μια πολύ καλή ομάδα και είναι βασική η παρουσία του Κοινοβουλίου. Πρέπει να ενισχύσουμε την δημοκρατική μας νομιμότητα στην Ιγυρία και είμαι στη διάθεσή σας εάν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Ντέλτσεβα έχει το λόγο τώρα. Ε, σε τέσσερα λεπτά τελικά, αντί για τρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να σε ευχαριστήσω και εγώ γιατί μου την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχα τιμή να προεδρεύσω και με τέσσερα μέλη εγώ, Τζιν Λάμπερτ ε, και ο Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρ και ο Μοντάλντο. Πήγαμε 13-18 Απριλίου στην Ιγυρία. Θα, θα ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τον ενθουσιασμό τους και την προσπάθειά τους, γιατί ακριβώς συμπεριφερθήκαμε πώς θα έπρεπε και εφερθήκαμε όπω θα έπρεπε. Να τους ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Πέτερλε, γιατί από την αρχή έτσι μας επέτρεψε να ενταχθούμε πλήρως στην αντιπροσωπή αυτή παρατήρηση. Ήταν πολύ καλή συνεργασία και παρατήρηση και έτσι μπορέσαμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να συντονίσουμε το μήνυμα το οποίο θελήσαμε να δώσουμε στη διάσκεψη στην ε, συνέντευξη τύπου και πίζα και την ομάδα της Γραμματείας του Κοινοβουλίου στην παρουσίαση του προγράμματος αντιπροσωπείας μας, ε, επίσης όμως και για τις συναντήσεις εκεί, συνομιλωτικές πολύτιμη βοήθεια, τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα το τίμημα, η πρόκληση αυτή. Είχαμε συναντήσεις κυρίως με τον καθηγητή Ζηγία και τον Good Luck Jonathan επίσης και με προσώπους της, της αντιπολίτευσης και από την κοινωνία των πολιτών ακριβώς σας τα λέω αυτά τα πράγματα γιατί σας δείχνει πως έχει κατάσταση ότι όλη αυτή η απόψή μας σχηματίστηκε και από τη βοήθεια των όλων των παρατηρητών. Να σας πω τι ακριβώς είδαμε επιτέλους και να ολοκληρώσουμε διάφορες συστάσεις ε, και μετά από τις παρατηρήσεις ε, στη μέρα των εκλογών ε, γιατί ακριβώς θα έχουμε εκεί μια έκθεση με περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ να σας πω ότι σχετικά με αυτές τις εκλογές, σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που συμφωνήσαμε όλοι, δεν ήταν ακριβώς όπως έπρεπε τουλάχιστον σε διεθνή πρότυπα να είναι αξιόπιστες και να έχουμε έτσι ε, να είναι κάτι το αξιόπιστο, το τίμιο και το πρώτο που παίχθηκε ήταν η αναβολή των εκλογών από τις 2 Απριλίου και μετά η διανομή του υλικού του εκλογικού και μετά αναβλήθηκαν οι εκλογές ακριβώς 9, 16 και 26 Απριλίου διαδοχικά. Να επιμείνω επίσης κάτι ότι για το εκλογικό σύστημα. Οι πρωτικές εκλογές βασίστηκαν σε μια ε, ειδική πλειοψηφία που έπρεπε ο καθένας τουλάχιστον στα δύο τρίτα των ε, κρατηδίων να έχει το ένα τέταρτο ψήφων τουλάχιστον. Αυτό λοιπόν σχετικά με την καταγραφή των υποψηφίων είχαμε 21 υποψηφίους ε, μία μόνο γυναίκα όμως, ε, να το σημειώσω αυτό, να το τονίσω αυτό. Και επίσης ε, είδαμε ο πρώην πρόεδρος που επέμενε να υποβαλεί και πάλι ψηφιότητα, υπήρξε αντίδραση, αλλά εδώ υπήρχαν Υπήρχε τέλο πάντων μια ενωμένη αντιπολίτευση και το είδαμε και τη μέρα πριν τι εκλογέ με μια τελευταία προσπάθεια για να μπορέσουν να κατεβούν μαζί και απέτυχε η προσπάθεια αυτή. Και εδώ να σα πω τι έγινε κατά τη διάρκεια τη εκλογή τη αλλά πρώτα απ' όλα έπρεπε να μείνουν ήρεμα τα πράγματα και να μην ασκηθεί βία. Τη μέρα των εκλογών ακριβώ είχαμε δύο ομάδε, στη Μπούζα και στη Μίνα, και να επιμείνω πάνω σε κάτι ότι το σύστημα το εκλογικό ε, πρώτα απ' όλα το πρωί μια πρώτη φάση και μετά ψηφορία τη δεύτερη φάση, ε, δηλαδή μια αναγνώριση των ψηφοφόρων την πρώτη φορά για να αποφύγουμε να ψηφίσουν αρκετές φορές κάποιοι και γι' αυτό μερικές φορές καθυστερήσαμε, υπήρξε ο κόσμος που αναγκάστηκε να κάνει ουρά, να γραφεί το πρωί και μετά να ξαναεπανέλθει το απόγευμα για να ψηφίσει. Οι εκλογές κατά γενικό τρόπο διεξήχθησαν ε, ήρεμα και μετάξυ και έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο το, το προσωπικό ασφαλείας που ήταν επαγγελματία πραγματικά και βοήθησαν πολύ επαναλαμβάνω. Τώρα εδώ να σας πω ότι τα πράγματα διέφεραν από την πόλη στην Ήπεθρο και ο συνάδελφος μπορεί να μας το επιβιώσει για μετά της ε, ρηφορία την εξεκλου... να σας πω τι έγινε. Κανείς ε, πριν από την επίσημη αναγγελία των αποτελεσμάτων δεν είπε ότι νίκησε κανεί υποψήφιο αντίθετα μα τι έγινε στην ε, ακτή του και αυτό ηρέμησε τα πράγματα. Και ε, από ό,τι είδαμε ο Τζόναθαν ε, ε, είχε εξελέγει από τη φορά και μετά ακούσαμε διάφορες πράξεις βίας αλλά η αντιπροσωπεία μας δεν ήταν αυτό από τις μάρτυρες παρόμοιων πράξεων βίας και μετά οι συστάσεις της αντιπροσωπείας μας αρκετά πράγματα πρώτα απ' όλα ενθαρρύνουμε την συμμετοχή γυναικών σε κάθε επίπεδο πολιτικής ζωής και ακόμα κάτι σχετικά με την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης και την ελεύθερη έκφραση θα πρέπει να ενισχυθεί, να τονωθεί και διάφορες βελτιώσεις που θα πρέπει να έχουμε για τον πλουραλισμό τον πολιτικό. Θα πρέπει η αντιπολίτευση να έχει τα μέσα για να υπάρχει και εκείνη και χρηματοδότηση της εκστρατείας ακριβώς. Θα πρέπει να προωθηθεί αυτό. Και ακόμα ένα σημείο σχετικά με τις εκλογές των νόμο του 2010. Ίσως θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε ακριβώς τι γίνεται σε περίπτωση διαμαρτυριών όταν παρεμβαίνουν τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών, των ψηφοφόρων και θα πρέπει να ενημερώνεται πάντα ο κατάλογος των ψηφοφόρων και επίσης τελευταίο σημείο για τα μέλη της ΕΝΙΚ που διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ε, να εγγυηθεί ακριβώς την ιδιωτερότητα, την αντικειμενικότητα αυτής της διαδικασίας της εκλογικής θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα αυτό και θα ήθελα να αναφέρω τα μέλη του σχεδίου Swift Count το 2011 ακριβώς με μια κατάλληλη διακασία, έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη οι πολίτες και εδώ και επίσης αυτό που θα δείκαμε εμείς, αυτό ακριβώς νιώσαμε, ε, περισσότερο καλύτερη ένταξη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επικεφαλής αντιπροσωπείας, αν ακριβώς έδειξαν σοβαρή στάση όλοι οι συνάδελφοι και έτσι και εγώ ίδια μπορώ να σας πω ότι μπορέσαμε πραγματικά να βοηθήσουμε για τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εκλογών αυτών στην Ιγυρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και η και τώρα το λόγο έχει Ευρωπαϊκή επιτροπή. Μελάντο. Ε, επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Μάλλον Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, από το τμήμα που ασχολείται με τον εκδημοκρατισμό και τις εκλογέ. Θα κάνω σύντομα σχόλια και θα δώσω το, δικαι... το... το λόγο στην συνάδελφό μου από την ίδια υπηρεσία που ασχολείται με, τα γεωγραφικά... Ε, με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η ε, Νιγηρία. Θα ήθελα να πω το εξή. Νομίζω ότι ήταν μια αποστολή παρατήρηση εκλογών πάρα πολύ επιτυχής, πολύ σημαντική για τις σχέσεις τη διμερή μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της Νιγηρία. Ε, ήταν μια αποστολή η οποία επέτρεψε την ενίσχυση του ρόλου και της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρου για την Ιγυρία, για την ε, εκλογική μεταρρύθμιση, για την μεταρρύθμιση της διακυβέρνηση, όπως επίσης για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της ε, σχέσης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νιγηρίας. Ήταν λοιπόν μια εκλογική παρατήρηση που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια σοβαρή επαγγελματική ε, ε, αξιολόγηση της όλης κατάστασης και έχει μια πολύ σημαντική και προστιθέμενη αξία στις διμερείς μας σχέσεις. Θα συνεχιστεί τώρα με την διατήρηση ε, της, ε, του δυναμικού αυτού που έχει δημιουργηθεί, ώστε να μην είναι μια απλώς, απλώς μια αποστολή παρατήρησης εκλογών, αλλά να είναι και να οδηγείς και στο επόμενο βήμα ε, των διμερών μας σχέσεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο στη συνάδελφό μου να μας πει περισσότερα. Η κυρία Μπράιτ. Η κυρία Μπράιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ε, από, την, ε, από την άποψη των γεωγραφικών δράσεων της ΕΙΕΔ πρόκειται για το συνδυασμό μιας έντονης περίοδη, περίοδου από το καλοκαίρι ήδη συνεργασίες και διαλόγου με, την, ε, με τις αρχές της Νιγηρίας και των όσων έπρεπε να γίνουν για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας με τη χώρα, οι μας με τη χώρα αυτή. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και είχαμε και ένα πολύ σημαντικό διάλογο στο πλαίσιο τριών ε, συναντήσεων ε, υπουργικού και ανωτάτων αξιωματούχων ε, με σκοπό την ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και τη βελτίωση της εκλογικής διαδικασίας στην Ιγυρία. Υπήρξαν κάποια, κάποιες πολλές θετικές ενδείξεις σε σχέση με την Ιγυρία. Ήταν σαφές ότι την Ιγυρία την απασχολούσε τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης ε, και τον αντίκτυπο και τα αποτελέσματα του αντικτύπου της Αραβικής Άνοιξης, όπως επίσης και το βαθμό ηρεμίας ε, που ήταν ε, ε, που κυριάρχησε στην μεγαλύτερη, κατά τη μεγαλύτερη περίοδο ε, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν βέβαια, υπήρξε κάποια αναστάτωση που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της, ε, των προεδρικών εκλογών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λάμπερτ. Θέλετε να απαντήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ. <clears throat> Πολύ χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω στην ε, αποστολή αυτή παρακολούθησης και θέλω να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Πέτερλε για τον πολύ ε, επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο διεξήχθη αυτή η παρακολούθηση και την στήριξη από το προσωπικό που υπήρξε ε, πολύ χρήσιμη. Ε, έχουμε επισημάνει διάφορες ανησυχίες, καταρχήν τα πλαίσια μέσα στα οποία γίνονται οι εκλογές. Είχαμε παρατηρητές σε ε, κάθε πλευρά, σε κάθε σημείο της Νιγηρίας και σε ορισμένες ορισμένες ε, περιοχές η έκβαση ήταν αμφισβητούμενη διότι η πολιτική κατάσταση στα ποτάμια, στο Δέλτα και τα λοιπά είναι δύσκολη και αυτό είναι ένα πολιτικό πρόγραμμα, πρόβλημα. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι η συμμετοχή ε, στις εκλογές ε, απέδειξε ότι θεωρούν πιο επουσιώδες είναι το ο κοινοβούλιο διότι τα πολλά λεφτά είναι αλλού στο πολιτικό σύστημα αλλά ήταν μία πρόκληση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουμε δηλαδή στη συνέχεια ε, τι συνέχεια δόθηκε στην αποστολή αυτή παρακολούθησης. Αν δηλαδή αυτό συνέβαλε για να υπάρξουν πιο στενές θέσεις με το Κοινοβούλιο της Νιγηρίας και μία βελτίωση των εκλογών. Γιατί πολλοί μας είπαν ότι οι εκλογές το 2011 είναι καλύτερες αλλά την επόμενη φορά θα πρέπει να έχουν βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι επαρκεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές ή πρέπει να εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας, δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε, είπαμε τα πάντα, πολύ καλά, υπέροχα μάλλον. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα. Αύριο το πρωί να σας ότι στην ίδια αίθουσα θα είμαστε και πάλι. Επίσης, ναι, στις 9 η ώρα. Και συνάδελφοι, παρακαλώ τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μην λησμονήσετε την κάρτα σας, έχει σημασία. Γεια σας, αύριο στις 9 το πρωί και πάλι.